Buonasera, abbiamo Καλό σα απόγευμα. Ξεκινάμε τι εργασίε μα. Περιμέναμε μερικά λεπτά προκειμένου να φτάσουν και οι καθυστερημένοι. Περνάμε στο πρώτο σημείο τη μισθή διατάξεω. Πρέπει να εγκρίνουμε το σχέδιο τη μισή διατάξεω. Έχει διανεμηθεί σε όλε τι γλώσσε και περιέχει την απαραίτητη τεκμηρίωση όλα, δηλαδή τα απαιτούμενα έγγραφα τώρα οι αναφορές που έχουν συμπεριφθεί σήμερα στη διάταξη σε πολλά σημεία θα εκπροσωπηθούν του αναφέροντες όπως η 6 για το αεροδρόμιο του, Βέτατς, του Σέφιλ, το 9 για το αεροδρόμιο του Βαράχας, υπάρχουν 13 για την Χιτά στην Ελλάδα, σημείο 16 και τα υπόλοιπα για τα δικαιώματα ιδιοκτησία στην Ιρλανδία και μετά οι, διατα... αναφορές για αύριο θα ασχοληθούμε με την οδική ασφάλεια στην Ιρλανδία και θα έχουμε παρόντα τον κύριο Φάρεν και τον κύριο Κίν. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε σε διάταξη. Περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Το δεύτερο σημείο αφορά στην έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεως της 14 Σεπτεμβρίου 2009. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά και αν ε, μέχρι το πέρας της συνεδριάσεως δεν υπάρχουν στάσεις από τα μέλη θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Ή μάλλον να στα εγκρίνουμε τώρα. Δεν βλέπω να υπάρχουν στάσει. Ε, μπορούν να εγκριθούν λοιπόν τα πρακτικά τη 14 Σεπτεμβρίου. Τρίτο σημείο τη μισή διατάξεω. Θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή πω ε, μετά από τη συνεδρία τη 19η Οκτωβρίου, όπου εξετάσαμε τις υποψηφιότητες για τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή, έστειλα τις επιστολές ε, στους ενδιαφερόμενους ε, για να τον ενημερώσω σχετικά με το ποιοι εγκρίθηκαν και ποιοι αποκλείστηκαν ε, εξάλλου. Έλαβα και τη γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας για το θέμα που έθεσε ο κ. Μπαρό, το οποίο βεβαιώνει όμω τα όσα είχε δηλωθεί προφορικά κατά τη διάρκεια τη Επιτροπή μα από την αρμόδια τη νομική υπηρεσία. Και αυτή η επιστολή θα διανεμηθεί. Έχει διανεμηθεί και ένα έγγραφο με προτώσει για το κλείσιμο ορισμένων ε, ε, αναφορών. Εάν δεν υπάρχουν στάσει, θα θεωρηθούν λοιπόν ότι εγκρίνονται οι αποφάσει ε, περί των αναφορών αυτών. Δεν ζητάει κανείς το λόγο. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο, σημείο 4. Che è il documento Συγγνώμη, περνάμε στο σημείο 5 που αφορά το έγγραφο εργασία για την ενική Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ένα χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη στην υπηρεσία των πολιτών, πρόγραμμα τη Στοχόλμη. Ε, η κυρία Βόλη ε, απουσιάζει για προσωπικού λόγου, αλλά εμεί θα πρέπει να περάσουμε στην έγκριση του εγγράφου, διότι το ψήφισμα θα ψηφιστεί την προσεχή εβδομάδα στις ε, τρεις ε, επιτυχίες αρμόδιες επιτροπές. Έχει διανεμηθεί σε όλους σας ε, το έγγραφο εργασίας για το χώρο ελευθερίας κλπ. Αλλά και οι τροπολογίες της κυρίας Βόλης που έχουν ήδη υποβληθεί τα βασικά σημεία που αναφέρονται στο έγγραφο εργασία ε, είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση, προσθέα ανηλίκων, συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμβέα αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η πολιτική θεώρηση ε, και το δικαίωμα διαμονή, ε, κοινωνικά δικαιώματα, συντάξει κλπ. Όσα άπτονται λοιπόν της ελεύθερη διακίνησης. Αυτά είναι σημεία τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο έγγραφο το οποίο μας απασχολεί, Λαμβάνεις υπόψη το χαρακτηριστικά των ζητημάτων αυτών που εξετάζει η Επιτροπή μας. Υπάρχει κάποιος που να επιθυμεί να λάβει το λόγο. Όχι. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία του κειμένου. Ψήφι υπέρ. Κοντράριο. Ψήφι κατά. Αποχές. Το έγγραφο έγινε δεκτό. Περνάμε τώρα στο τμήμα Α, Αναφορέ προσυζήτηση. συζήτηση. Η πρώτη αναφορά είναι 505.008 του κ. Στίο Ντάλτον, Βρετανού υπηκόου, που αφορά τη διαμετρία κατά των σχεδίων για το κλείσιμο του αερολιμένα του Σέφιλντ. Ο αναφέρον είναι παρόν και θα ήθελα να δώσω το λόγο. Καλησπέρα σα. Τον ε, Οκτώβριο του 1998 θεωρήθηκε ότι η πόλη μου, η πόλη του Σέλφιλτ, θα έπρεπε να είχε το δικό της αεροδρόμιο. Γιατί ε, θα ήταν διαφορετικά μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ε, πόλεις χωρίς αεροδρόμιο. Αποφασίστηκε λοιπόν να δημιουργηθεί ο παρέτος οργανισμός για να κατασκευάσει το αεροδρόμιο αυτό, το οποίο θα πήγε 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, θα ήταν προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς και επίσης προβλεπόντουσαν ότι οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα για τη μεταφορά μέχρι το αεροδρόμιο αυτό θα ήταν πολύ χαμηλότερες από ό,τι μεταφορά για άλλα αεροδρόμια. Επίσης, το αεροδρόμιο αυτό θα κάλυπτε 32 εκτάρια, τα οποία δόθηκαν στους, ε, στον οργανισμό κατασκευής του αεροδρομίου αυτού που θα γινόταν με ε, δημόσια χρηματοδότηση. Για ένα τμήμα του αεροδρομίου αυτού δόθηκε μάλιστα και κοινοτική χρηματοδότηση. Από τη στιγμή που δόθηκε η απόφαση για την κατασκευή του αεροδρομίου αυτού, ετέθηκε η προπόθεση ότι το αεροδρόμιο θα έκλεινε μόνο αν, αν αποδεικνυόταν εμπορικά ζημιογόνο. Μετά όμως από την πάροδο μόνο τεσσάρων ετών, η αρμόδια κατασκευάστρια επιχείρηση Peel Holdings, που έχει επίσης δημιουργήσει και το αεροδρόμιο Finengley για την Βρετανική πολεμική αεροπορία, αποφάσισε να αγοράσει το Sheffield City Airport. Δόθηκαν τότε οι απαραίτητες εγγύσεις ότι θα συνεχιζόταν φυσιολογικά η ε, εκμετάλλευση του νέου αυτού αεροδρομίου και με κάποιες αλλαγές που έγιναν στη συνέχεια από την ε, εταιρεία αυτή. Υποβαθμίστηκε η ε, κατηγοριοποίηση του αεροδρομίου όσον αφορά την ασφάλεια από την κατηγορία 5 προς την κατηγορία 3 με αποτέλεσμα να μειωθεί η κίνηση στο αεροδρόμιο αυτό και να καταστεί τελικά το αεροδρόμιο λιγότερο ανταγωνιστικό. Τους επόμενους 12 μήνες πάρα πολλά τερματικά τμήματα του αεροδρομίου μετατράπηκαν σε γραφεία. Επίσης, ε, το σύστημα ε, προσγείωσης ILS σταμάτησε να χρησιμοποιείται συστηματικά. Θελήσαμε παρόλα αυτά να διατηρήσουμε το αεροδρόμιο όσο πιο λειτουργικό γίνεται και να καταφέρουμε να ε, εγγυηθούμε τις προδιαγραφές ασφάλειας του αεροδρομίου για περίοδο 10 ετών προκειμένου να δικαιολογηθεί η απόφαση για, για το πρώιμο αυτό κλείσιμο του αεροδρομίου, δόθηκε ένα αυτόνομα ανεξάρτητο έγγραφο προς τις αρμόδιες αρχές, το οποίο είχε πάρα πολλά λάθη. Λεγόταν, για παράδειγμα, ότι ε, θα χρονόταν κάποια μίσθωση για το αεροδρόμιο αυτό, το οποίο θα συνέβαινε μόνο αν ε, το αεροδρόμιο αυτό ε, είχε αποδειχθεί τελικά ότι ήταν οικονομικά βιώσιμο. Επίσης φάνηκε ότι δεν είχαν γίνει οι απαραίτητε επιχορηγήσει για το αεροδρόμιο. Αυτό θα θέλαμε λοιπόν από την Επιτροπή να εξετάσει τα ακόλουθα σημεία. Γίναν οι απαραίτητε προσπάθειε προκειμένου να καταφέρουμε να προσελκύσουμε επιχειρήσει προ το αεροδρόμιο αυτό και τελικά διατηρήθηκε το αεροδρόμιο αυτό σε τέτοιε συνθήκε προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσω από τι αεροπορικέ γραμμέ. Δεύτερον, ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι το αεροδρόμιο δεν είχε κανένα μέλλον και ότι όλε οι λειτουργίε του αεροδρομίου αυτού θα μπορούσαν να μεταμεθωθούν στο νέο αεροδρόμιο της εταιρείας Πύλη στο Φίνιγκλεϊ. Και τρίτο ερώτημα, πώς θα μπορούσε ένα αεροδρόμιο να είναι οικονομικά μη βιώσιμο την στιγμή που είχε χρεωθεί το ποσό των 297.000 λίρων για τη λειτουργία του. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να σας πούμε ότι Ορισμένες, ε, ορισμένοι προορισμοί, για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Πολωνία, εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο του Σέφιλτ και ακολουθούνται όλες οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη λειτουργία του αεροδρομίου αυτού. Επίσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η οικονομία του Σέφιλτ είναι χαμηλότερη από ό,τι προβλέπεται στον μέσο όρο του Ηνωμένου Βασιλείου για πόλεις ανάλογου μεγέθους. Επομένως υπάρχει ένα έλλειμμα της τάξης του 1,1 δισεκατομμυρίου λιρών που θα πρέπει πιστεύουμε να καλυφθεί και θα μπορούσε στην κατάσταση αυτή, στην βελτίωση μάλλον αυτή να συνεισφέρει το νέο αεροδρόμιο. Ζητάμε από την Επιτροπή να συνειδητοποιήσει ότι κανεί από του αναφέροντε δεν έχει κάποιο οικονομικό συμφέρον μέσω τη αναφορά αυτή. Βρισκόμαστε στην αίθουσα αυτή γιατί πιστεύουμε ότι χάνουμε μια πολύ σημαντική υποδομή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την οικονομική βιωσιμότητα τη πόλη μα. Ο μόνος ο οποίος ε, βγαίνει τελικά κερδισμένος από την όλη αυτή η ιστορία είναι ο εργολάβος ο οποίος θα εκμεταλλευτεί αυτό το νέο χώρο. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια δημόσια ανοιχτή διερεύνηση για το τι ακριβώς ε, συνέβη, για το πώς αποφασίστηκε το κλείσιμο και η πώληση του αεροδρομίου. Το λιγότερο μπορούμε να στήσουμε αυτή τη στιγμή είναι όλες οι δημόσιες δαπάνες που επενδύθηκαν για την κατασκευή του αεροδρομίου αυτού να επιστραφούν από τους εργολάβους που ανέλαβαν την κατασκευή του αεροδρομίου. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, κύριο Δίξον. Thank you, Chairman. The... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απάντηση είναι πολύ σύντομη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία εξουσία προκειμένου να αποφασίσει τον διατήρηση ενός αεροδρομίου ή το να ανοίξει ένα αεροδρόμιο, να κλείσει ένα αεροδρόμιο κλπ. Αυτό εντύπτει στην ε, τοπική, σε τοπική πρωτοβουλία. Αυτό το οποίο μπορούμε να επιδώσουμε είναι ότι το αεροδρόμιο είναι κλειστό από το 2002. Δεν είχε ποτέ πολλές προγραμματισμένες πτήσεις. Το πιο κοντινό αεροδρόμιο έγινε σε απόσταση 46 χιλιόμετρων από το Σέφιλντ και από διακινεί 1,5 εκατομμύριο επιβάτες ετησίως. Το, ένα, επόμενο, το επόμενο αεροδρόμιο είναι το Μάντσεστερ, το οποίο εξυπηρετεί 22 εκατομμύρια επιβάτες, βρίσκεται σε 90 χιλιόμετρων από το Σέφιλντ και η διαδρομή απαιτεί ένα, μία ώρα και 15 λεπτά. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι τα όσα έχουν φασίσει για το Σέφιλντ ε, είναι σύμφωνα με τα όσα έχουν φασίσει και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κίρκοφ έχει λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον αναφέροντα για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε την υπόθεση αυτή απογοητεύτηκα πάρα πολύ από την απάντηση της Κομισιόν. Εγώ είμαι ε, για το Γιώργο και Χάμερ και τέως ε, εκφέφωνο για τα θέματα μεταφορών για, την, για το κόμμα μου. Είμαι επίσης ένα επίτιμο μέλος της Ένωσης ε, ε πιλότων στο Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ ίδιος ε, έχω την άδεια πιλότου. Τα λέω αυτά γιατί ήθελα να ξέρετε ότι έχουν εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά τα θέματα, εδώ και πολλά χρόνια. Είδα μάλιστα η Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν για τα περιφερειακά θέματα τότε να έχουν πολύ κατανάλωση και είπανε ότι συζητάμε για ένα σημαντικό ποσό δημοσίων πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηριχθεί μια εμπορική εκμετάλλευση που όπως είπε ο αναφέρον δεν έχει ακολουθήσει καθόλου μια γραμμή ευθύνη, ε, βασιζόμενο ακριβώ σε αυτό το θέμα της χρηματοδότηση τη οποία έτυχαν. Είναι νομίζω ότι και να πούμε, κύριε Πρόεδρε. Ότι δεν εξετάζουμε το θέμα των εμπορικών αναπτύξεων, εγώ καταδικάζω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σέφιλ. Νομίζω ότι η Γενική Διεύθυνση Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει πώς έχουν ταπανηθούν τα χρήματα αυτά. Και επίσης, ε, θα ήθελα να μου απαντήσει και το, τοπικό, το συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με αυτή την έκθεση που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη. Καθόλου ανεξάρτητη δεν είναι και μια που πρόκειται για σημαντικά ποσά, είναι ένα θέμα που είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν ζητάει από την Κομισιόν να αρχεί να διοικεί αεροδρόμια. Πολλά έχουν να κάνουν. Είναι απλώς να αναλάβουν τις ευθύνε τους, ώστε χρήματα που έχουν δαπατηθεί και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά δικαιούται το Νότιο Ιόξαρ επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν. Αλλά το τι γίνονται τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα η Κομισιόν και η Αρμόδιοι να κάνει τις απαραίτητες έρευνες όπως ζήτησαν οι αναφέροντες, να εξεταστεί το θέμα προσεκτικά και αν έχει γίνει κάτι το εσφαλμένο μέχρι στιγμή σε οποιοδήποτε επίπεδο θα πρέπει να διορθωθεί κατάλληλα. Περιτέρω φαίνεται εντυπωσιακό Και μάλιστα ήθελα να σας πω ότι αυτό, αυτό το αεροδρόμιο Robin Hood και θα σας πω ότι ο Robin Hood είναι από το Nottingham και το αεροδρόμιο είναι στο Yorkshire που αποκρίνεται. Τέλος πάντων φαίνεται σαν να γίνεται μια επικάλυψη. Και τα δύο αεροδρόμια είναι στο νότιο Yorkshire και πολύ κοντά. Και πιο κοντά από ό,τι ανέφερε η Κομισιόν. Δεν ξέρω πού κοίταξαν. Αλλά στο Exeter είχαμε μια παρόμοια υπόθεση. Και είχε πει η Κομισιόν τότε ότι δύο αεροδρόμια που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και πάρα πολύ κοντά το ένα στον άλλο δεν μπορούν να ανήκουν στον ίδιο εκμεταλλευόμενο. Και τώρα εγώ δεν θα σταματήσω να εξετάζω την υπόθεση. Πραγματικά ε, δεν μπορώ παρά να συγχαρώ τους αναφερνούς για τον ευγενικό και γενναιόδωρο τρόπο με τον οποίο ε, έχουν αντιμετωπίσει το θέμα και δεν ήταν καθόλου ε, ικανοποιητική η απάντηση που εδώ. Uh, um, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη από τους αναφέροντες γιατί δεν ήμουν παρόν όταν ε, παρουσίασαν την ε, αναφορά τους αυτή. Του ζητώ λοιπόν συγγνώμη. Ωστόσο πρέπει να πω ότι γνωρίζω την υπόθεση αναφοράς αυτής διότι ε, έχει φτάσει ήδη από το 2008, δηλαδή από την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής Αναφορών, τον ήμουν μάλιστα και την πρόεδρος Επιτροπής αυτής. Σε καμία περίπτωση δεν διαφωνώ με τα όσα είπε ο κύριο Κέρκοπ στην ε, παρέμβασή του, με τον οποίο συνεργάζομαι και σε άλλη επιτροπή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, θα ήθελα να πω το ακόλουθο. Αν υπάρχουν αποδείξεις ότι η αξιολόγηση αυτή που έλαβε χώρα δεν ήταν ανεξάρτητη, τότε θα μπορούσαμε κι εμείς να την έχουμε και θα μπορούσε η Επιτροπή να λάβει τα στοιχεία αυτά, τις αποδείξεις αυτές, γιατί μόνο βάσει των αποδείξεων αυτών μπορεί είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων, όχι των εθνικών πόρων. Μιλάμε εδώ για κοινοτικούς πόρους. Και εμείς στη συνέχεια θα μπορούσαμε να λάβουμε μία απόφαση για το αν μπορούμε να πιστέψουμε τα πορίσματα αυτή της ανεξάρτητης αξιολόγησης. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους αναφέροντες και από τον κύριο Κέρκοπ να μας δώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις που θα αποδεικνύουν τελικά ότι αυτή η ανεξάρτητη αξιολόγηση δεν ήταν τελικά ανεξάρτητη. Και να πω και κάτι ακόμα. Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή σαν νομοθέτες, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα θα έλεγα. Από τη μια λέμε ότι θέλουμε οι πολίτες να ταξιδεύουν ελεύθερα, να φτάνουν γρήγορα στα αεροδρόμια, να μπορούν να πάνε στην Κώστα Ντελσόλη, στην Ιταλική Ριβιέρα, εύκολα και γρήγορα, αλλά την ίδια στιγμή ως νομοθέτες πρέπει να εξορροπήσουμε το ζήτημα αυτό με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, με την εκπομπή διοξιδίων του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου. Η απόφαση λοιπόν για το κλείσιμο ενός αεροδρομίου θα πρέπει να ληφθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από τους ε, ιδιοκτήτες του αεροδρομίου αυτού. Συνεπώς υφίσταται το δίλημα αυτό. Είμαι σίγουρος όμως ότι ο κύριος Κέρκοπ θα συμφωνήσει μαζί μου όταν λέω το εξής. Αν ένας φορέας είναι ζημιογόνος, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι για να τον κρατήσουν εν ζωή. Αυτά είχα να πω για ένα ζήτημα, για μια αναφορά που θεωρώ την ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί πάρα πολλά στοιχεία της αναφοράς αυτής βασίζονται σε ε, αιτιάσεις, χωρίς να έχουμε όμως κάποιες πραγματικές αποδείξεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν τις αποδείξεις αυτές και παράλληλα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι προωθούμε σαφώς τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά παράλληλα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον αναφέροντα και τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Είμαι σε θέση να πω πως η συντομία δεν είναι πάντα προτέρεμα, ακόμα στους Κομισιόν μα είχε αναγγείλει ότι η παρέμβασή του θα είναι σύντομη, αλλά αυτή η σύντομη παρέμβασή του δεν νομίζω πω ε, επέφερε την προσδοκούμενη απάντηση που εμεί ε, θέλαμε να λάβουμε. Είναι κάτι το οποίο επανέρχεται συχνά στην Επιτροπή μας και αφορά τη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που κανένα όψή μας ε, δεν μπορεί να βλέπει αδιάφορους τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, του εκτελεστικού. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε εδώ την λόγο αναφορά και πως είναι σαφές ε, το αίτημα το οποίο προέκυψε από τις παρεμβάσεις των αδέλφων για μια περαιτέρω εμβάθυνση του ζητήματος ο πλευράς Κομισιόν, ε, πως εξάλλου ανέφερε και ο αναφέρον εμείς λοιπόν ως Επιτροπή θα θέλαμε να προωθήσουμε κάποιο αίτημα αποσαφήνισης και από την Επιτροπή Προπολογισμών. Θα ήθελα να προσθέσω πως ε, η Επιτροπή ζήτησε για περαιτέρω στοιχεία από τον αναφέροντα προκειμένου να βοηθήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην, ε, στις ερευνές της Ναι, αναφίβολα και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Νομίζω λοιπόν πως ε, αυτά μπορούν να είναι συμπερέσματα μας τώρα. Αν αναφέρουν θέλει να προσθέσει κάτι, κάποιο νέο στοιχείο, του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ που εξετάζετε την ε, αναφορά μας. Ε, ευχαρίστως θα σας διαβιβάσουμε ένα αντίγραφο της όλης υπόθεσης που αφορά στο αεροδρόμιο του Σέφιλντ. Έχουμε επίσης και έναν κατάλογο περίπου 100 σημείων που αφορούν σφάλματα που έχουν διαπιστωθεί. Ευχαρίστω λοιπόν να τα διαβάσουμε σε εσά ή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη αναφορά. Αναφέρον είναι ο κύριο Μάρκο Νέβης Σίλβα, Πορτογαλική Ιταγένεια, ο οποίο όμω δεν παρίσταται, δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ευρωπή Αρνάν Δελεσκρίλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από την υποβολή της αναφοράς, ο αναφέρον υπέβαλε δύο επιστολές στην Κομισιόν του 2006 σχετικά με το αεροδρόμιο του Πόρτο. Η Κομισιόν το έλεγε πάρα πολύ σοβαρά και απάντησε στις ε, επιστολές αυτές και ζήτησε μια αντίδραση από τις πορτογαλικές αρχές για να διορθωθούν τα σφάλματα που υπάρχουν στο αεροδρόμιο του Πόρτο. Οι πορτογαλικές αρχές ήταν συνεργάσιμες και υιοθέτησαν κάποια συμπληρωματικά μέτρα ο αναφέρον ενημερώθηκε σχετικά. Δεν ικανοποιήθηκε γιατί δεν ενωθήθηκαν ένομα μέσα κατά των πορτογαλικών αρχών. Και κατά τη γνώμη του η αντίδραση δεν ήταν αρκετά γρήγορη. Να υπάρχει μια απάντηση μέσα στο 2006. και υπέβαλε μαζί με την αναφορά του και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με ε, εικαζόμενες παρεμβιάσεις ασφαλείας Ρολουμένα παράκταση της Μαδρίτης. Η Κομισιόν απάντησε λέγοντας ότι το 2006 και το 2007 διαβεβαιώθηκε με τις τοπικές αρχές ότι έχουν επιληθεί τα προβλήματα που παρουσιάζει ο αναφέρον. και είπαμε τα κρατημένα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και, <clears throat> η Κομισιόν κάνει μια επιθεώρηση. απλώ. Όταν υπάρχουν ελλείψεις, η Κομισιόν εξασφαλίζει την διόρθωσή του. Αν δεν λάβει χώρα μια διόρθωση των λήψεων αυτών, η Κομισιόν εκείνη τη δικασία επί παραβάση κατά του εν λόγω κράτους. Από το 2004 μέχρι σήμερα η Κομισιόν έκανε πάνω από 100 επιθεωρήσεις αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγιναν και 50 στο επίπεδο πρώτων μελών. Από τις τελευταίες παρατηρήσεις που σας στείλαμε εδώ, έκανε η Κομισιόν και μία επιθεώρηση και του Μαδρίτη Παράχας και του Πόρτο. Και οι δύο αυτοί είδαμε ότι δεν έχουν πια τα προβλήματα που είχε αναφέρει ο αναφέρον. Και το 2008 ο αναφέρον υπέβαλε μία αίτηση για να δει όλα τα εν λόγω έγγραφα. Η Κομισιόν ορίθηκε όμως να του στείλει τις επιστολές που είχε ανταλλάξει με τα κράτη-μέλη, γιατί αυτή θεωρείται ότι είναι ε, απόρριτη ε, ε, ενημέρωση σύμφωνα με το κανονισμό 1049. Τα υπάλληλα στοιχεία του τα είχαμε δώσει. Και όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε δώσει τα έγγραφα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιτρουγκάιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εν συντομία να πω ότι υπάρχουν παράξενες περιπτώσεις. Εδώ αναφέρον ε, ε, μιλάει για διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης για να δει κανείς αν μπορεί να περάσει κάποιο κουτάκι κοακόλας από κάποια σχισμή ε, αν πληρούνται όλε όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας κλπ. Νομίζω πως η Κομισιόν ήταν ξεκάθαρη και με τις ερωτήσεις που έκανα και τις οποίες, και απαντήθηκα και αναφέρονται εδώ στον ίδιο φάκελο που έχετε και εσείς αναχείραστο, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα πως πρόκειται για μια αναφορά η οποία αφισβητήθηκε και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να την κλείσουμε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένο με τις απαντήσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Τροπή. Αυτά. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις υπάρχουν. Εντάξει. Μπορούμε να κλείσουμε την λόγο αναφορά. Όλοι ικανοποιημένοι. Πάμε παρακάτω. Περνάμε στην αναφορά υπερθμών 8 του κ. Άξελ Μπάντο, γερμανική σταγένεια, σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τα σχόλια της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα. Βάσει της ε, έκθεσης που εστάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, το αεροδρόμιο του Σένεφελτ δεν θεωρείται μείζον αεροδρόμιο σύμφωνα με την οδηγία. Σύμφωνα με την οδηγία του 2007, τα επίπεδα θορύβου θα πρέπει να εξολογούνται βάσει των στοιχείων που υφίστανται για το προηγούμενο έτος, στη συγκεκριμένη περίπτωση του 2006 λαμβάνονται υπόψη οι μετακινήσεις που γίνανε στο Σόνενφέλτ 50.000 για το 2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια έκανε μία ανάλυση των, του θορύμπου, που ε, η, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη και Στη συνέχεια ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη τον Ιούλιο του 2009 να μας αποστείλουν τα περαιτέρω στοιχεία. Ζητήθηκε από τη Γερμανία να, αποστάλει, να αποστείλει με συγχωρείτε, περαιτέρω στοιχεία για το αεροδρόμιο του Σόνεφερ. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει την απαραίτητη δράση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων που στείλαν τα κράτη-μέλη στο τέλος δηλαδή του έτους ή στις αρχές του 2010. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την απάντησή της. Μπορούμε όμω ε, να αναρωθούμε το εξής. Έχουμε τα τα μέσα στη διάθεσή μας ε, προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση που επικρατεί στο ε, ζήτημα του θορύβου, το θέμα τη συγχωρήπανσης. Σύμφωνα από ό,τι γνωρίζω, υπολογίζουμε, υπάρχουν κάποιοι, ε, κάποιοι κανόνες, κάποιοι πίνακες, ε, αλλά αυτό τι σημαίνει. Υπάρχει και πρέπει νομοθεσία για να διασφαλίσει πως η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω. Αυτό το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε εδώ είναι ότι οι άνθρωποι υποφέρουν από αυτήν την ρήπανση μπορούμε να καταγράψουμε την, ε, ε, τη δυσαρέσκεια αυτή των ε, ανθρώπων, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε αυτή την ηχορύπανση, έχουμε κάποια νομοθεσία, κάποιο εργαλείο κατάλληλο προκειμένου να εφαρμοστεί μια πιο αυστηρή νομοθεσία, ιδιαίτερα στις χώρες που έχουν μια νομοθεσία ανεπαρκή επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τουργκάτη, έχει το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στην Επιτροπή. Αν κατάλαβα καλά, η Κομισιόν ζήτησε στοιχεία και δεν, στα οποία δεν απάντησε όμως το κράτος μέλος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μιλάμε για μια αναφορά η οποία εστάρει το 2007. Έτσι δεν είναι κυρία Πρόεδρε. Το 2007 λοιπόν ζητήθηκε στην Γερμανία να ενημερώσει την ε, Επιτροπή για το γεγονός αυτό και δεν έλαβε ούτε μία απάντηση. Εμείς ε, λάβαμε λοιπόν την ε, αναφορά αυτή και στείλαμε και μία επιστολή στην ε, Γερμανία λέγοντάς ότι εδώ και δύο χρόνια σας έχει έχει γίνει η αναφορά αυτή και δυστυχώς ε, δεν μας έχετε ενημερώσει και δεν μπορούμε να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας έναν Ευρωπαίο πολίτη διότι δεν ε, μας ενημέρωσε το εμπλεκόμενο κράτος μέλος. Λοιπόν, δύο χρόνια όπως καταλαβαίνετε είναι πολλής χρόνος, ε, δεν είναι δυνατόν να μην πρόλαβα να απαντήσουν και δυστυχώ εδώ σήμερα εμεί δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τον Ευρωπαίο αυτόν πολίτη. Θα ζητούσα λοιπόν να αφήσουμε εκκρεμή την αναφορά αυτή και να ζητήσουμε στη γερμανική κυβέρνηση να απαντήσει και έτσι η Κομισιόν να μπορέσει με τη σειρά της να απαντήσει στην αναφορά του ενδιαφορομένου. Ο της Κομισιόν θέλει να προσθέσει κάτι ή να απαντήσει ενδεχομένω. Σας ευχαριστώ. Άκουσα τις παρατηρήσεις που γίνανε να απαντήσω στην πρώτη. Η οδηγία όσο έχει αυτή τη στιγμή λέει ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν για τις ωραϊκές τιμές του ρήβου. Βάσει λοιπόν της υφιστάμενης νομοθεσίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα κατά κράτους μέλους αν ε, υπερβαίνονται σε κάποια περίπτωση τα όρια θορύβου τα οποία τίθενται, όπω σα είπα, από την Εθνική Νομοθεσία. Από την άλλη, όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί την ε, υφιστάμενη οδηγία. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία και περιμένουμε ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε μια νέα πρόταση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο του 2011. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν διαδικασία αναθεώρηση οδηγία. Εξετάζουμε πολλέ πτυχέ οδηγία αυτή με του απαραίτητου εμπειρογνώμονε, με του αρμόδιου εμπειρογνώμονε και εξελίσσεται ακόμα αυτή η εργασία. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη παρατήρηση. Συμφωνώ ότι η αναφορά αυτή υποβλήθηκε πριν από αρκετά χρόνια. Ωστόσο, τους ε, χάρτες θορύβου δεν τους λάβαμε όλους μαζί. Τα κράτη-μέλη αποστήλαν τους χάρτες θορύβου με διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε ως έγγραφα, άλλοτε με email και μετά την ε, προθεσμία του 2008. Και μετά λάβαμε και κάποιες αναθωρημένες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Προκειμένου να αξιολογήσουμε τα, τους χάρτες θορύβου, χρειαζόμαστε τουλάχιστον έξι μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενο των χαρτών αυτών. Θα πρέπει να μεταφραστούν όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται εκεί και συνέχεια καλούμεθα να αξιολογήσουμε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στους χάρτες θορύβου. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε κατά οριζόντιο τρόπο να λάβει δράση βάσει της αξιολόγησης που περιλαμβάνει βάσει εξολόγηση που έγινε του, των χαρτών θορύβου και φέτο είμαστε πλέον σε θέση να δούμε αν θα πρέπει για κάποια κρατημέλη να κινήσουμε τη διαδικασία επί παραβάση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Καταλάβαμε πως ε, και η Κομισιόν επιθυμεί να αφήσει σε κρεμότητα την αναφορά αυτή προκειμένου να φτάσουν ε, οι απαντήσεις. Περνάμε τώρα στην υπαριθμό 9 του Μάρκ Σόουερ, Βιλική Σταγένεια, ε, συνοδευόμενη από 8 ακόμα υπογραφέ. Δώσω το λόγο λοιπόν στον αναφέροντα. Καλησπέρα σας. Έχω βρει μια μικρή παρουσίαση, αν θέλετε, με διαφάνειες. Λοιπόν, αγαπητοί μέλη της Επιτροπής, ε, θα ήθελα καταρχήν να σας παρουσιαστώ. Λέγομαι Μάρκα Ντεσαόρη και ζω στο Τρεις Κάντος, μια πόλη βόρεια-δυτικά από το αεροδρόμιο της Μαδρίσης. Ο λόγος που είμαι εδώ είναι ότι σε 7 Ιουλίου 2005 οι Ισπανικές Αρχές εισήγαγαν νέες ε, διόδους ε, εξόδου από το αεροδρόμιο της Μαντρίσης. Μία από αυτή ήταν η Radial 322 που άνοιξε σε ένα φυσικό δρυμό. Και το Φεβρουάριο του 2006 είχε αυξηθεί η συγκοινωνία σε 300 αεροπλάνα ανά ημέρα. Και αυτό οφείλεται σε ένα τέταρτο διάδρομο, λέγεται επίσημα. Αλλά δεν είναι αληθές αυτό. Το θέμα είναι ότι οι αρχές απελευθέρωσαν μεγάλα τμήματα των εδαφών εκεί που χρησιμοποιούνται τώρα για κατοικίες, δηλαδή για να κατασκευαστούν μάλλον κατοικίες. Βλέπετε εδώ διάφορα παραδείγματα, το Πράτο Νόρτε στην Αλγέντε, μετά η Φέντα Λούκα και η Ντέζα Βιέχα. Επίσης έκλεισαν οι αρχές την δίωδο Ναβασκόρτας πάνω από ένα ε, μεγάλο στρατιωτικό ε, πεδίο εκπαίδευσης που λέγεται Ελγκολόσο το νέο αυτό, η νέα αυτή ιδιότητα στο Radio 322 περνάει από μια περιοχή προστασίας, ε, φυσικό, φυσικής προστασίας του τεινών, συγγνώμη, που ανέει Σότο Ντεβινιουέλας. Και βλέπετε εδώ ποια, γιατί προστατεύεται από το Natura 2000, από το UNESCO Biosphere Reserve, το Special Area for Protected Birds ε, και η ε, σημαντική περιοχή για πουλιά και Community Interest Site. Αυτό τώρα υπάρχουν, εκεί υπάρχουν διάφορα πτηνά που βλέπετε που είναι ε, χαρακτηρισμένα ως ε, ε, δέοντα ειδική προστασίας. Υπάρχουν επίσης ζώα όπως κάποια ελάφια που είναι επίσης προστασέφημα. Τι δεν έκαναν οι αρχές. Οι αρχές πριν αρχινήξουν το Radial 322 δεν έκαναν μία έρευνα περιβαλλοντολογική για την δίωδο αυτή. Μόνο γύρω από το αεροδρόμιο έκαναν την έρευνα αυτή. Η τελευταία αξιολόγηση είναι από το 1999 και καλύπτει τα αρχικά, τις αρχικές ε, διόδους που υπήρχαν πριν από το 2005. Επίσης, δεν ζητήθηκε καθόλου η άποψη των πολιτών. Και αυτό τι σημαίνει τελικά ότι με υψηλά επίπεδα θορύβου καταδικάζονται ε, περιβαλλοντικά προστατεύσιμες περιφέρειες. Η, ο θόρυβος είναι πάνω από 80 δεσιμπέλ. Υπάρχουν επίσης περισσότερα δυστυχήματα ε, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα κολέγιο 1500 φοιτητών εκεί από κάτω. Και τέλος, οι επιπτώσεις για τους κατοίκους είναι πάρα πολύ σημαντικές που κατοικούν στο Τρεσκάντος, στο Σεμπαστιάν Τελορέγες και αλλού. Αυτό τι σημαίνει, ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι Ισπανικές θέσεις καταπατούν την οδηγία για το περιβάλλον 92 κάθετος 93, 97 κάθετος 62 και 85 337, την οδηγία για την προστασία των πτηνών 79 409 και την Οδηγία Συμμετοχή των Πολιτών 2003-35. Και έχουμε και κάποιες πολύ τελευταίες ε, πληροφορίες. 7 Μαου τρέχοντο, οι αρχές τη είχαν μια αλλαγή. Το 80% των αεροπλάνων πετά την αποχείωση γυρίζουν στο δεξιά προς τα βόρεια. Και γι' αυτό γιατί οι πόλεις του Τρεσκάντο και του Κολμένα Φιέχο προωθούν δύο νέες ε, ε, δύο νέους οικισμούς με, με 7.000 διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται οι ισπανικές αρχές για τους νέους οικισμούς οικονομικά παρά για την προσοχή του περιβάλλοντος και των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, πιεστούν οι Ισπανικές αρχές να κλείσουν το Radial 322 και τα αεροπλάνα να ακολουθούν τις διόδους που υπήρχαν πριν από το 2005, όπως υποστηρίζεται αυτό και από περιβαλλοντικές μελέτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να δώσω το λόγο στον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριο Τζαντονόβιτς, ε, ή κάπως έτσι. Εκπροσωπώ την ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Λάβαμε αρκετές πληροφορίες σχετικά με την αναφορά αυτή. Έχουν αναλυθεί οι πληροφορίες αυτές και σε σχέση με τους ε, διαδρόμους ε, Radial 322 πάνω από την περιοχή Σότο Ντεβίνιο που αποτελεί τμήμα του Natura 2000. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί προς την Επιτροπή δεν μας επιτρέπουν να κρίνουμε ότι αυτός, αυτή η παρενόχληση είναι σημαντική σε ό,τι φορά την ε, προστασία αυτής της ε, περιοχής. Και έτσι σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 4 ε, κάθετος 3 για τον Σικοτόπους και την προσία της άρης πανέσης χλωρίδας η Κομισιόν δεν θεωρεί ότι η, η βλάβη για την φανή και τη χλωρίδα στην περιοχή είναι υψηλή. Σημειώσαμε αυτά που είπε ο αναφέρον. Κράτησαμε τα στοιχεία που ανέφερε στην παρουσίασή του, αλλά τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα στη θέσή μας δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε, <clears throat> στο συμπέρασμα ότι παραβιάζεται η κοινοτική οδηγία σχετικά με αυτόν τον ε, αεροδιάδρομο. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω <clears throat> να παραμείνει ανοιχτή η λόγω αναφορά και να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια νέα έκθεση και να ζητήσει στις Ισπανικές αρχές, ειδικά στην ΑΕΝΑ που είναι και υπεύθυνη για αυτούς τους αεροδιαδρόμους το αεροδρόμιο των Μπαράχας, εάν γίνεται σωστή χρήση των ρυθμίσεων που αναφασιστεί αναφορικά με τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις των αεροσκαφών. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τις Ισπανικές αρχές τα κατάλληλα στοιχεία για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να απαντήσουμε στους ε, αναφέροντες. Είναι πολύ σημαντική η αναφορά κατά την άποψή μου Θέλουμε να λάβουμε περαιτέρω προφορίες από την Κομισιόν και δεύτερον να ζητήσουμε να τηρούνται οι κανόνες γύρω από το αεροδρόμιο Μπαράχας προκειμένου να μην υπάρχει πλέον η χορύπανση και να περιορίσουμε την ζημιά τόσο στην Πανίδα Χλωρίδα αλλά και στους γύρω κατοίκους περιοχές. Ο αναφέρον θέλει να προσθέσει κάτι. No, thank you for listening to me. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Πρόεδρος, συμφωνώ με το αίτημα του συναδέλφου να παραμείνει ανοιχτή η υπόθεση για να ζητήσουμε περαιτέρω προφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ γενικόλογη η απάντησή της προς το παρόν. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια περαιτέρω επαλήθευση των καταγγελιών διότι διαβάζοντας ε, τα έγγραφα μας δίνεται η εντύπωση ότι δεν έχει βαθυνθεί το ζήτημα από την Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν περαιτέρω επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις ε, και συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Στο σημείο αυτό μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση επί της αναφοράς μεν, αλλά το θέμα παραμένει, παραμένει σε εκκρεμότητα. Περνάμε στην επόμενη αναφορά, είναι παριθμόν 10 του κ. Κόντραντ Βαζνιεύσκη, Πολωνική Σταγένεια, σχετικά με το σχέδιο κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα διασχίζει προστατευόμενη περιοχή βορειοδυτικά τη παρσοβία Δίνω τον λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην εκπρόσωπο, μάλλον, κ. Τσάντονοβιτ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αναφορά αυτή έχει να κάνει με έναν δρόμο στα βόρειο-δυτικά της Βαρσοβίας, ένα αυτοκινητόδρομο ουσιαστικά, που θα δημιουργηθεί ανάμεσα σε δύο οικοτόπους που υπάγονται στην περιοχή Natura 2000. Οι πολωνικές αρχές κάνανε μία αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου και στη φάση αυτή έχουν δώσει μια περιβαλλοντική άδεια όσον αφορά μια προτινόμενη διαδρομή για την κατασκευή αυτού του αυτοκινητόδρομου. Κατά την άποψή μας λοιπόν οι πολωνικές αρχές κάναν τη δουλειά τους, εξέτασαν δηλαδή την, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που θα έχει το σχέδιο αυτό για το Natura 2000 και για τις δύο προτινόμενες διαδρομές που βρίσκονται κοντά στους δύο αυτούς οικοτόπους και επέλεξαν τελικά την λύση εκείνη που θεωρείται ότι είναι η λιγότερο ζημιογόνος για το περιβάλλον, βάσει των προδιαγραφών του Natura 2000. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι αρχές της Πολωνίας έκαναν το καθήκον τους και δεν υπάρχει κανένας λόγος να διερευνήσουμε περισσότερο, να αφισβητήσουμε τις αποφάσεις που έλαβαν. Η τελική όμως άδεια κατασκευής για τον αυτοκινητόδρομο αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει δοθεί θα ακολουθήσει ακόμα μία διαδικασία περαιτέρω αξιολόγησης, όπου θα πρέπει να εξεταστούν και οι τεχνολογικές τεχνικές λύσεις για την κατασκευή του δρόμου αυτού, να ληφθούν υπόψη και οι χάρτες θορύβου, οι διαδρομές που ακολουθούν ορισμένα ζώα τα οποία μετακινούνται στην περιοχή αυτή και στη συνέχεια μετά την αξιολόγηση αυτή θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παροχή της άδειας κατασκευής. Αυτό προβλέπεται για τον Νοέμβριο του 2010. Με τα δεδομένα όμω που ισχύουν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι πολιτικέ αρχέ δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του. Κάνανε την περιβαλλοντική μελέτη που έπρεπε να γίνει για τι περιοχέ Natura 2000 και από ό,τι φαίνεται ο δρόμος αυτός πρέπει αναγκαστικά να περάσει κοντά στις δύο, στους δύο αυτούς οικοτόπους Natura 2000. Γίνανε όλες οι απαραίτητες αναλύσεις και μολονότι λάβαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον αφέροντα, δεν μπορούμε εμεί να θεωρήσουμε ότι οι πολωνικέ αρχέ δεν κάνουν σωστά το καθήκον του ή δεν προχώρησαν σε όλε τι περιβαλλοντικέ εξολογίε που πρέπει να κάνουν στα πλαίσια του Natura 2000. Επιθυμεί να λάβει κάποιο το λόγο. Επειδή δεν παρίσταται ούτε ο αναφέρον, μπορούμε να θεωρήσουμε επαρκής ε, της ε, εξηγής της Κομισιόν και να θεωρήσουμε πως κλείνει στο σημείο αυτό η αναφορά. Περνάμε στην επόμενη αναφορά, την υπαριθμόν 11, κρύου Κάρλο Ολντάνη και άλλων 5 Ιταλών ε, για την παράκαψη του πάρκου στο Τιτσίνο και του Γεωργικού Πάρκου νότιος του Μιλάνου αναφορικά με εντηρήσει για το σχέδιο υποδομή αυτοκινητοδρόμου που παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τι παραγωγικέ επιπτώσει για τη διαφάνεια δημοσίων έργων. Δεν παρίσταται ο αναφέρον. Η Λάουρα Ταμπελίνη εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά έχει γίνει ήδη αντικείμενο επανειλημμένων ανακοινώσεων προς το Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες περαιτέρω προφορίες ε, που μας είχε ζητήσει ο αναφέρον 12 Ιουνίου. Ο αναφέρον αναφέρει ότι, τα, ότι το σχέδιο έχει προοδεύσει και σύμφωνα με τον αναφέροντα ε, οδηγίες 85-37 δεν ε, τηρούνται και η οδηγία 92-43 η ονομαζόμενη ε, οδηγία για τους οικοτόπους. Ζήτησε λοιπόν πέντε επιφορές από τις Ιταλικές αρχές σχετικά με την ε, έλεγχο της, ε, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων η Κομισιόν θα συνεχίσει να ενημερώνει την ε, Επιτροπή σας σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της ε, έρευνας ε, που διεξάγει. Διευθύνουν οι Ιταλικές Αρχές. Ευχαριστώ. Παραμένει ανοιχτό το θέμα. Περνάμε την επόμενη αναφορά στο σημείο 12 της μεσαίας διατάξεως του κ. Κόσμου Φρακάσου, Ιταλικής Ταγένειας, σχετικά με την ανησυχία για τις διοξίνες στο Τάραντο να δώσω το λόγο ξανά στην Λάουρα Ταμπελίνη. Ευχαριστώ. Όπω αναφέρεται ήδη στην γραπτή απάντηση προ την Κοινοβουλία, η Κομισιόν είναι σε επαφή με τι Ιταλικέ Αρχέ για να ε, έχει τι πληροφορίε για την 9661 την λεγόμενη IPPC οδηγία. 2008-1 για την επιχείρηση Ήλβα στην οποία αναφέρεται ο αναφέρον. Η απάντηση που δόθηκε από τις αλληλικές αρχές επιβεβαιώνει ότι πραγματικά αυτή η οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί. Από την άλλη μεριά όμως η εν λόγω κατάσταση δεν είναι σύμφωνη με την οδηγία και είναι σε αντίθεση με το άρθρο 5.1 που προβλέπει πλήρη συμμόρφωση μέχρι 30 Οκτωβρίου 2007. Οι ιταλικές απαντήσεις δείχνουν επίσης ότι το πρόβλημα είναι πιο διευρυμένο στο ιταλικό επίπεδο. Μια διαδικασία επιπαραβάση για την οδηγία EPPC ξεκίνησε ήδη και σύμφωνα με τις τελευταίες απαντήσεις ε, των Ιταλικών αρχών δεικνύουν ότι οι άδειε βάση του IPBC δεν έχουν ακόμα δοθεί για διάφορους λόγους και γι' αυτό στις 2 Φεβρουαρίου 2009 γνωμοδότησε η Κομισιόν και η Κομισιόν απάντησε τον οι Ιταλικές Αρχές συγγνώμη, απάντησαν τον Απρίλιο του 2009. Η Επιτροπή θα σας κρατήσει ενήμερους για οποιοδήποτε εξελίξεις θα υπάρχουν προσεχώς. Σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω ότι είναι πολύ ο χρόνος ε, για μια ρήπανση η οποία μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες ε, επί των υγείας των πολιτών. Αν θα μπορούσε λοιπόν η Κομισιόν να επιταχύνει κάπως την όλη διαδικασία και να απαντήσουν έγκαιρα οι Ιταλικές αρχές, διότι πρόκειται για μια αναφορά η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Πρόεδρος. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια αναφορά η οποία υποβλήθηκε το 2007 και αν ε, πράγματι υπήρχε κάποιος συναγερμός, ε, κάποια ιδιαίτερα ψηλή ανησυχία, θα είχαμε ήδη θύματα. Εν η Κομισιόν παρακαλώ να επιταχύνει τι διαδικασίες και να φροντίσει να λάβει απαντήσεις έγκαιρος Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη αναφορά. Με ενημερώνουν πως ε, για την αναφορά στο σημείο 13 δεν ε, παρίσταται εκπρόσωπος της Κομισιόν ακόμα. Περνάμε στην αναφορά βρίσκεται στο σημείο 14 της Νέας Διατάξεως, ε, έχει υποβάλει ο κ. Ντέισμέ, Ιρλανδική Σταγέννη Ξεώμη της Western Hill Fisherman Association, σχετικά με τον αποκλεισμό των αλλιών από διαδικασία κατάρτιση του προγράμματος διαχείρισης του χελιού στην Αλδιά. Μπρέντα Νόσε, έχει το λόγο, εκπρόσωπος Κομισιόν. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα και με την λόγο λόγω αναφορά, του 14. Στο σημείο αυτό. Δεν έχουμε πρόσωπο ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 14. Ο κύριος Αρμάνο Γκονζάλες παρίσταται για το σημείο 15. Ούτε. Δεν παρεμπίσκεται ο κύριος Σαρμάν. Για να πάμε παρακάτω να δούμε τι θα γίνει. Δουλέψαμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαν προβλέψει οι υπηρεσίες και έχουμε προχωρήσει στις αναφορές που είχαν προβλεφθεί για τις 16 και 25. Μήπως κατά τύχη βρίσκεται κάποιος εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Τροπή για τις ε, επόμενες αναφορές. Όχι. Στο σημείο αυτό δεν μας απομένει παρά να διακόψουμε τις εργασίες μας για λίγα λεπτά. Μέχρι ότου... Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Άρτια αφιχθήσα η κυρία. μερικά να προλάβει να ανασάνει. Ε, θα ξεκουραστούμε για 10 λεπτά περιμένοντας όλους τους εκπροσώπους από όλες τις υπόλοιπες αναφορές. Ε, επομένως ε, μπορείτε να πάρετε λίγο χρόνο και θα τα ξαναπούμε σε 10 λεπτά. Ε, δεν χτύπησα εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε. <laughs> Ευχαριστώ τον κύριο Λόπ που το έκανε. Ε, πάμε λοιπόν στην αναφορά αριθμός 13 και έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, βελγικής ε, τον αναφέροντα. Ε, η αναφορά σχετίζεται με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Ελλάδα. Ε, κύριε Παπαδόπουλο, μπορείτε να παρουσιάσετε την αναφορά σας. Ε, θα μιλήσω γαλλικά. C'est plus facile pour moi de parler en français. Είναι πιο εύκολο για μένα να μιλήσω στα γαλλικά. Κυρίε και κύριοι μέλη τη Επιτροπή Αναφορών, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εξ των Επιτροπών για την καταπίεση ε, τη πραγματοποίηση των εγκαταστάσεων στο, Καρβουνάνη και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μα δίνετε τη δυνατότητα να σα εκφραστούμε εδώ γιατί είσαστε οι μόνοι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδίδετε ιδιαίτερη σημασία στο φάκελό μας. Από τότε που ανησυχούμε για το περιβαλλοντικό έγκλημα μέχρι τη μέρα που είμαι εδώ μπροστά σας σήμερα δηλαδή έχει περάσει πάρα πολλού χρόνο. Δυστυχώ το καρβουνάρι όπως προβλέπετε τα ύδατα του ποταμού ήδη έχουν ε, έχουν μολυνθεί από τα λεγόμενα λιξιβιάτ. Την ημέρα στην οποία έγραψα την αναφορά αυτή, κάτω από την εντύπωση της σύγκρουσης μου με αστυνομικούς ρομπότ, δεν ήξερα τι είναι μια υγειονομική ταφή, μια ευρωπαϊκή οδηγία, ε, μελέτη ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. Εν τω μεταξύ όμως μελέτησα το θέμα, τη γεωλογία, της ε, ε, τους χώρους υγειονομικής ταφής, ε, μελέτησα τις οδηγίες, τους κανονισμούς και ενημερώθηκα σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με τους φίλους μου, το Λευκή, το Ελληνικό και το Γραμματικό, ταχθήκαμε κατά τους μεθόδου που ακολουθείτε στην Ελλάδα και θα σας δώσω πολλά στοιχεία για να καταλάβετε τι γίνεται και στο Καρβουνάρι αλλά και στη Λευκήμη και αλλού. Όσον αφορά τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την λόγω οδηγία 85337, οι μελέτες αυτές, παρόλο το υψηλότατο κόστος τους, δεκάδων χιλιάδων ευρώ, είναι γεμάτες με ανακριβείς στοιχεία, βασίζονται σε στοιχεία από την ε, βιβλιογραφία και δεν βασίζονται σε μετρήσεις επιτόπου. Το 2009, το μάη του 2009, πολύ διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες μίλησαν για μια ε, βιομηχανία ελληνική ελληνική paste για τις μελέτες αυτές. μας χάνει. στο καρβουνάρι λέγεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς πήγαμε στην περιοδομία, πήραμε τα σχέδια του χωριού και είδαμε δύο εκπλήξεις. Δηλαδή ότι η πραγματική απόσταση ε, ανάμεσα στα όρια του καρβουναριού και ε, ε, του χώρου ταφής είναι 131,51 μέτρα. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Αυτοί που έκαναν τη μελέτη και πληρώθηκαν δεκάδες χιλιάδων ευρώ δεν ενημερώθηκαν καν βάσει των επισήμων χάρτων της πολιοδομίας. Ούτε μέτρησαν τίποτα ήδη επί τόπου. Η ανάλογη μελέτη της Λευκήμη παραβλέπει την ύπαρξη δύο ποταμών που βρίσκονται σε 190 και 340 μέτρα από τον χώρο της ταφής αυτής και δεν αφαίνεται καθόλου στις ε, τουριστικές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις σε λιγότερο από 500 μέτρα. Οι δύο μελέτες αυτές παράβλεψαν τις σημαντικές δραστηριότητες ε, εκτροφής ζώων ακριβώς που συνορεύουν με τις, τους χώρους αυτούς ταφής. Πώς μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε τις μελέτες αυτές αξιόπιστες που σας έδωσα τόσο απλά παραδείγματα για το ότι δεν είναι πραγματικά βάσιμες. Και πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε έτσι τις ε, αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όσον αφορά τη 1991 κάθος 31 και τη 2006 κάθος 12, έχω να πω ότι η συγγραμματοδότηση των χώρων υγειονομικής ταφής από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται σε ειδικού όρους που προβλέπουν το να υπάρχει μια δομή για την διαλογή, την ανακύκλωση και την αξιολόγηση των απορριμμάτων πριν να ταφούν. Αλλά ούτε στο καρβουνάρι ούτε στη λευκή υπάρχει τέτοια ε, δομή στους ε, τόπους αυτούς υγειονομικής ταφής πάνε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Από την άλλη μεριά, η... ο χώρος ταφής του Καρουνάρη λειτουργεί από την 12η Πρώτου 2009 χωρίς άδεια των αρμοδίων αρχών. Η του του νομού της Θεσπρωτείας ζήτησε μάλιστα να σταματήσει η λειτουργία από 13 Φεβρουαρίου 2009 ευτυχώς σταμάτησε επιτέλους η λειτουργία της βάσει της λαϊκής κατακραυγής. Στο φάκελο που θα σας δώσω όταν τελειώσει η παρουσίασή μου έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία ότι εδόθησαν άδειες χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 10 χρόνια μέσα συγχρηματοδότησε δύο χώρους υγειονομικής ταφής στη Θεσπροσία για να καλυφθεί η Θεσπρωτεία και η Πρέβεζα. Αλλά όπως βλέπετε η μία από αυτές η Κοριτιανή δεν λειτουργήσε ποτέ. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν παντού χωματερές ε, αχαλήνοτες και ανεξέλεγκτες. Γιατί πολλές από τις ε, τοπικές αυτοδιοίκησεις δεν θέλουν να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους τόσο μακριά. Όπως παραδείγματο χάρη ή η Γουμενίτσα που εξακολουθεί να ρίχνει τα απορρίμματά της στην Καστρίνη, μία ανεξέλεκτη χωματερή. Κατόπιν έρχομαι στη 2006 κάθος 60, 2008 κάθος 1 και έχω να πω ότι πραγματοποιώντα ε, τους χώρους αυτούς αυτή του Γραβουνά τη Λευκήμη, η, το ελληνικό κράτος υποτίθεται ότι προστατεύει το περιβάλλον, ενώ ακριβώς ο τόπος, ε, ο οποίο έχει επιληφθεί για τους χώρους αυτούς είναι αντίθετος με οποιοδήποτε έννοια της προστασία του περιβάλλοντο. Τα το βλέπουμε αυτό από την κακή λειτουργία στο καρβουνάρι όπου έχουμε αποδεκτικά στοιχεία ότι τα απόβλητα αυτά λίματα, τα λήξια βιάτ, πέφτουν σε μία κοιλάδα που είναι του ποταμού Κοκκίτος που καταλήγει στον Αχέροντα που έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο βάση του Natura 2000. Βλέπετε τα στοιχεία αυτά που σας παρουσίασα σε αυτή τη διαφάνεια που είναι μπροστά σας. Άμα θέλετε θα σας δώσω εγώ το σχετικό βίντεο για να δείτε πραγματικά πώς κινούνται αυτά τα λίμματα. Βλέπετε να εκεί είναι αυτός ο όγωγος που πάει στο ποτάμι κοκκίτου αυτό που κάνανε για, προστατευτικό, για να προστατεύσουν κάπως είναι ότι σταματήσαν να, να τραβάνε πόσιμο νερό από το προδρόμι. Βλέπετε εδώ. Βλέπετε πού είναι αυτή η εγκατάσταση της, του χώρου υγειονομικής ταφής και είχαμε εδώ αυτό το σημείο για το πόσιμο είδο που έχει κλείσει τώρα και που θεωρήθηκε σαν το πιο ε, χαρακτηριστικό στοιχείο το ότι έχει κλείσει για να μπορέσει να γίνει εκεί. Και ε, θα μπορούσαν αλλιώ να έχουν επιλέξει να, να έχουν επιλέξει την ε, τοποθεσία ανατολικά του καρβουναριού. Καταλαβαίνετε, κλείνουμε τη γεώτρωση και τελείωσε. Και υπάρχουν και χειρότερα. Στη Λευκήμη όταν έσκαψαν γη το Μάρτιο-Απρίλιο 2008, κατακλήθηκε όλος ο χώρος από νερό, γλυκό νερό, καλό νερό και έγινε μια λίμνη. Σταμάτησαν λοιπόν οι εργασίες λόγω της πλημμύρας αυτής. Η εμπειρογνωμοσύνη που ζητήθηκε και που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο γεωλογικών ε, και ορεικτών ερευνών ανεξάρτητου οργανισμού που υπογράφεται από τον κύριο Ζαχαριουδιάκη αποδείχθηκε ότι πρόκειται για ε, νερό, για ένα υδροφόρο, υδροφόρο στρώμα που επικοινωνεί με όλα τα σημεία τροφοδότησης ύδατος γύρω-τριγύρω και γι' αυτό είπε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να εγκατασταθεί ο χώρος αυτός υγειονομικής ταφής ακριβώς εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένας δεν θέλησε να σεβαστεί το περιβάλλον για να κάνει κάποιες οικονομίες χρημάτων. Βλέπετε εκεί στον άραχθο, τον άραχθο στον οποίο ε, κατεβαίνουν όλα αυτά τα λίματα κατευθείαν λίματα και πετρέλαια. Το ίδιο γίνεται και στο γραμματικό. Να, σας το δείχνω εδώ. Έχουμε και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, δεν θέλω όμως τώρα να τα αναπτύξω όλα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω εδώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Μαρία Κουλούρη, μια μητέρα σαν δύο ετών που σκοτώθηκε από την επίθεση των ε, οργάνων τάξης που προσπαθούσαν να επιτρέψουν στους μπουλντόζες να περάσουν για να φτάσουν στη Λευκήμη. Εν κατακλείδη, θα σας δώσω μία σειρά α, επισήμων εγγράφων, βίντεο και φωτογραφιών που αποδεικνύουν αυτά που σας λέω. Εμείς πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από τον παραλυσμό μεταξύ των ε, εγκαταστάσεων του Καρβουνάρη, Λευκήμη Γραμματικό και στο Ελληνικό, αλλά όχι όμως αν ξέρετε ότι οι μελέτες έγιναν από τις ίδιες εταιρείε. Δηλαδή ΕΠΕΜΑΕ για το καρβουνά ελληνικό, Φραντζής ΕΠΕ για τη Λευκήμη και Ευρωπλάν ΕΠΕΜ Φραντζής για το γραμματικό. Στην πρώτη απάντηση που πήρα από εσά, απάντησα με περισσότερες ε, λεπτομέρειες και με περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για τα εγκλήματα αυτά. Και τέλος υπέβαλα την ε, αναφορά μου σε 2009 καθώς 4306. Δύο φορές ε, με δέχτηκαν και με άκουσαν ε, υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος. Και πραγματικά είδα ότι ήταν πολλοί από αυτούς Έλληνες. Θα ήθελα να μην ε, ξεχνάμε ότι δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρήματα, από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν δεκάδες σύλληψεις ή η μόνη εγγύηση για την αντικειμενικότητα που έχουμε εμείς είναι αυτή η αναφορά εδώ. Δεν ήρθα όμως για να ζητιανεύσω τη βοήθειά σας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήθελα για να προασπίσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταδείξω ότι υπάρχει ένα κράτος που καταποπατά τις ευθύνες που έχει αναλάβει. Επίτηδες, εγνώση του. Αυτά όλα καταδεικνύουν ότι η επιλογή αυτών των ε, τοποθεσιών ήταν ένα σφάλμα προγραμματισμένο και οργανωμένο για να περιοριστεί το κόστος ε, της ε, ταφής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ειλικρινά, μετά από 5-10 χρόνια θα δώσετε εσείς στα παιδιά σας λάδια από ή κρέας από το καρβουνάρι. Αλλά ξέρω επίσης σήμερα καλύτερα τι θα πει αναφορά και τι θα πει οδηγία. Και σας παρακαλώ να γίνουν σεβαστές οι οδηγίες 85 337, 1999 31, 2006 12, 2006 60 και επίσης 2008 1 και η εφαρμογή όλων των κυρώσεων που προβλέπεται από τις εν λόγω οδηγίες. Θα ήθελα επίσης να ε, αναγνωριστεί το σφάλμα εκτίμησης που έκανε η Ελλάδα κάνοντας την επιλογή για το Καρβουνάρι και Λευκίνη και τους άλλους φακέλους για το ελληνικό και το γραμματικό και να σταματήσουν αμέσως η χρήση του καρβουναριού. Σας παρακαλώ να ασκήσετε κυρίες βουλευτέ την απαραίτητη πίεση για νέα προγραμματισμό στην Ελλάδα βασιζόμενη σε πραγματική επιστημονική εργασία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ε, η κυρία Θα μιλήσω αγγλικά. Γνωρίζουμε το πρόβλημα αυτό στο καρβουνάρι. Ο αναφέρον πολύ σωστά είπε ότι εδώ πέρα έχουμε καταγράψει μια περίπτωση παράβασης. Ήρθαμε σε επαφή με τις ε, ελληνικές αρχές Λάβαμε πρόσφατα και την απάντησή τους, θα πρέπει όμως να αξιολογηθεί πρώτα με όλους πιθανούς τρόπους και υπό το φως της αρμόδιας οδηγίας στην οποία αναφέρθηκε ο αναφέρον. Επίσης, οι συναδελφοί μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδρίασαν τον Οκτώβριο παρουσία του αναφέροντος και άλλων αναφέροντων για το ζήτημα αυτό. Του ζητήθηκε τότε αν είχαν περαιτέρω πληροφορίες να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του φακέλου αυτού. Και μέχρι στιγμής λοιπόν αξιολογούμε τις διαθέσιμες πληροφορίες τόσο στα πλαίσια των ε, καταγγελιών και στα πλαίσια των απαντήσεων που μας έχουν δώσει οι ελληνικές αρχές. Ε, υπάρχει κάποια ερώτηση από μέρους του ακροτηρίου, του συναδέλφους. Κυρία Σας ευχαριστώ. Από το 2008 έχουμε την ε, αναφορά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο καιρό θα κρατήσει ακόμα την αναφορά αυτή ανοιχτή και μάλιστα τη στιγμή που δεν έχουμε μια πραγματική απάντηση. Η υπόθεση είναι δύσκολη γιατί ε, εσείς μας δώσατε αρκετά στοιχεία Φαντάζομαι ότι η Επιτροπή της έλαβε, δόθηκαν ε, κάποιες απαντήσεις από τις ελληνικές αρχές και από ό,τι φαίνεται το ζήτημα δεν προχωρεί. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι μιλάμε εδώ πέρα για χώρους υγειονομικής ταφής. Ξέρετε ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει τα πάντα. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε περιοχές πλούσιες σε νερό με πολύ σημαντικές για τις καλλιέργειες οι χώροι αυτή η υγειονομική σταφή είναι απαραίτητη, είναι σημαντική, Κανεί όμω δεν, του δεν τους θέλει δίπλα του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πιέσουμε τι ελληνικέ αρχέ να δώσουν γρήγορα μια απάντηση, προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση και να τοποθετηθούν οι χωματερέ αυτέ στο καλύτερο δυνατό σημείο. Και είναι σημαντικό να ληφθεί υπέψη ο παράγοντα περιβάλλον, γιατί αυτό που τελικά μα απασχολεί, είναι τι πλανήτη θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μα και στα εγγόνια μα. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, και στη Γαλλία είχαμε τα ίδια προβλήματα και φαντάζομαι ότι ανάλογα προβλήματα έχουν εντοπιστεί και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε απαντήσεις γρήγορα. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε. Ναι, ο κύριο Γιάννη. Ja, zum, äh, zum äh, möchte ich nur... Καταρχήν χαίρομαι που η Κομισιόν καταλήγει τώρα σε διαφορετικό συμπέρασμα από τις 27 Δεκάτου όπου έλεγε ότι όλα είναι θαυμάσια, όλα είναι εντάξει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί είναι πάντα αυτό το πρόβλημα, δηλαδή. Άλλο είναι αυτό που υπάρχει επί χάρτου. Θεωρώ ότι τα έγγραφα έχουν υποβληθεί σωστά κλπ. Από την άλλη μεριά έχουμε την πραγματικότητα όμως. Θα ήθελα λοιπόν να παρακολουθήσω την Κομισιόν να μην βασιστεί μόνο στο χαρτί, να βασιστεί στην πραγματικότητα. Να γίνει μια επιτόπου επιθεώρηση και αν βέβαια αποδειχθεί ότι είναι σωστό αυτό που ακούσαμε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνει. τι, είναι, τι να σας πω, δεν θέλω να πω απάτη, αλλά πάντως δεν είναι τα πράγματα έτσι ξεκάθαρα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υποβάλλονται κάποια έγγραφα και μετά λένε εντάξει θα κάνουμε μετά ό,τι θέλουμε εμείς. Θα ήθελα λοιπόν να εξετάσει η Κομισιόν λίγο και το θέμα των ανεξελέγκτων χωματερών. γιατί κανένας πραγματικά όταν κινείται στην Ευρώπη συλλέγει κάποιες εντυπώσεις. Αυτό είναι ένα σημείο που με απασχολεί και εμένα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέπτη, Μία ερώτηση θέλω να κάνω στην εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θα ήθελα να μας θυμίσει, αν είναι εύκολο, ε, πότε ακριβώς δόθηκε απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση και με δύο λόγια τι λέει η απάντηση αυτή τη κυβέρνηση, η οποία βεβαίω στο μεταξύ έχει αλλάξει, έχουν γίνει εκλογέ και έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Δυστυχώς ε, δεν μπορώ να είμαι πολύ ακριβή στην απάντησή μου όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ωστόσο βέβαια η αναφορά κατεγράφει την άνοιξη τρέχοντος αμέσως έγινε μια κοινοποίηση προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές και στη συνέχεια η απάντηση από τις αρχές αυτές πρέπει να έφτασε κάποια στιγμή το καλοκαίρι, στο τέλος του καλοκαιριού. Εδώ και δύο μήνες πάνω κάτω έχουμε την απάντησή τους. Όσον αφορά το περιεχόμενο της απάντησης αυτής, Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες, ε, διότι δεν ασχολούμαι άμεσα με την υπόθεση αυτή. Επειδή έχει να κάνει όμω με πάρα πολλές τοποθεσίε που αναφέρονται και από τον αναφέρονται, αλλά και με άλλα μέρη που καλύπτονται ε, από το ίδιο ζήτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση στο στομότερο δυνατό αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι μας έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες. Να ενημερώσω ότι ε, στάλθηκε μια απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση στις 25 Σεπτεμβρίου του 2009 ε, την οποία επεξεργάζεται από ό,τι καταλαβαίνω η Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσω στο, στους συναδέλφους ότι παρά την αμηχανία την οποία αισθάνομαι δεδομένου ότι ε, ε, η Μελίδα το καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο πράγμα ευχαριστώ τον κύριο Παπαδόπουλο ότι έφερε στο προσκήνιο μια τόσο δύσκολη υπόθεση. Ε, να υπενθυμίσω ότι η καινούργια κυβέρνηση της στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε θέματα περιβάλλοντος και ε, ε, ε πράσινης ανάπτυξης γενικότερα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει άμεσα αντίδραση. Ε, εμείς μπορούμε ως Επιτροπή να στείλουμε μια δεύτερη επιστολή με το συγκεκριμένο θέμα στην ε, ελληνική κυβέρνηση, στο καινούργιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και δεν θα απέκλεια καθόλου την δυνατότητα, εφόσον συμφωνούν τα μέλη της Επιτροπής, να πάμε στην, ε, να, να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα πάει να δει επί την ε, κατάσταση και να βγάλει τα συμπεράσματά της αν θεωρείται ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είστε για την ε, Επιτροπή, όχι. Εκτός αν η μετάφραση δεν ήταν καλή. Would you like to have a, a fact-finding committee visiting the site? Συμφωνείτε να συσταθεί μια διερευνητική επιτροπή που θα πάει επί τόπου. Solve it in the, with the coordinators. Do you agree? Συμφωνείτε, ωραία. Okay. Okay, then. Ε, κύριε Παπαδόπουλο, έχετε να προσθέσετε κάτι? Euh, euh, Αναφερόμενο στην ε, συνάδελφό σα, είπε ότι κανεί δεν θέλει να έχει λίματα στον κήπο του. Ναι, μα ακριβώ αυτό όμω έγινε στο καρβουνάρι. Όχι μόνο φτάσαν στον κήπο μα τα λίματα, αλλά στο σαλόνι μα. Το καρβουνάρι είναι ένα με, μια περιοχή που αποδέχθηκε τελικά να δημιουργηθεί ένα χώρο υγειονομική ταφή και ενώ αρχικά προβλεπόταν ε, μία απόσταση αποδεκτή από, τον, ε, από το χωριό αυτό, από την περιοχή αυτή. Ο φορέας κατασκευής την έφερε πολύ πιο κοντά. Εμείς ουσιαστικά στο Καρβουνάρ δεν ε, έχουμε τη στάση αυτή η οποία αναφέρθηκε από τη συνάδελφο, ότι δεν θέλουμε καθόλου να έχουμε στον κήπο μας μια χωματερή. Εμείς αποδεχθήκαμε να γίνει κάτι τέτοιο. κυρία Οσέα. Ο κύριος Οσέα. Οσί. Οσί. Οσί. Οκ. I'm here to respond to the e θα ήθελα να απαντήσω στην αναφορά που έχει γίνει για το χέλι, για τη διαχείριση του χελιού. Ε, με τον κύριο Ντι Μέι, Ιρλανδικής Ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Western Eel Fishermen Association και ισχυρίζεται ότι έχουν αποκλειστεί οι αλληλείς από τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος διαχείρισης του χελιού για την Ιρλανδία. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να απαντήσω στην αφορά του κυρίου Ντεσμέη όσον αφορά την κατάρτιση προγράμματος διαχείρισης του χελιού για την Ιρλανδία και που άπτει ουσιαστικά του κανονισμού 1100 κάθετος 2007. Μολονότι οι αλείς χελιών, οι βασικοί ενδιαφερόμενοι, τελικά συμμετείχαν στη δικασία σχεδιασμού μόνο στα τελευταία στάδια, όταν ήταν δυνατές αλλαγές, όταν ήταν δυνατές ελάχιστες μόνο πλέον αλλαγές. Σύμφωνα με τον αφέροντα, το πρόγραμμα που υποβλήθηκε είναι μεροληπτικό σε ό,τι αφορά τη δομή, τα πορίσματα και τη μέθοδο και δεν αντικατοπτρίζει απόψει κοινότητα των αλλιών χελιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα όσα λένε οι εκπρόσωποι των αλλιών χελιών και αυτό φαίνεται και στο άρθρο 2, 2 της κοινή αλληλευτική πολιτική. Δηλαδή, λαμβάνουμε πάρα πολύ, σημα... πάρα πολύ σημαντικά υπόψη την διαβούλευση με του ενδιαφερόμενου. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου του 2005, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση όσον αφορά την ανάκτηση των αποθεμάτων χελιού. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, στη συνέχεια, ο κανονισμός 1100-2007 του Συμβουλίου κατέρτισε τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκτηση των αποθεμάτων του Ευρωπαϊκού Χελιού. Θα ήθελα να πιστεύω στην προσοχή σας στο ότι η Ιρλανδία είχε ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία μιας εθνικής ομάδας εργασίας για τη διαχείριση του χελιού προτού εγκριθεί ο κανονισμός Συμβουλίου. Είχε δηλαδή ήδη από το 2006 το δικό της εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης χελιού. Στο πλαίσιο αυτής της Εθνικής Ομάδας Εργασίας, το Μάρτιο του 2008, επεστάλλει μία ενημέρωση προς εμάς από την αρμόδια εθνική αρχή της Ιρλανδίας, όπου λεγόταν, γινόταν λόγος για την πολύ άσχημη κατάσταση των αποθεμάτων χελιού. Ξεκίνησε συνέχεια μια διαβούλευση από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2008 και εκπροσωπήθηκαν όλοι οι λιμένες όπου δραστηριοποιούνται αλλοίς χελιών. Είχαμε έντονη συμμετοχή εκ των οποίων, και η σημαντικότερη συμμετοχή ήταν από τους αλλοίς χελιών. Όντως και αυτοί αναγνώριζαν ότι ε, τα αποθέματα χελιού βρίσκονται σε πολύ δεινή κατάσταση τα στοιχεία αυτά λήφθησαν υπόψη από τι ομάδε εργασία σε εθνικό επίπεδο και τα μέτρα τα οποία πρότειναν οι αλλοί δεν θεωρήθηκαν ε, επαρκή προκειμένου να ανακτηθούν τα αποθέματα χελιού και να επανέλθουν στα αποδεκτά τους επίπεδα. Γίνανε και απαραίτητες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες ε, επιβεβαίωσαν δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο με τα μέτρα τα οποία πρότειναν οι αλείς. Στη συνέχεια μετά την έγκριση της, του κανονισμού του Συμβουλίου, η Ιρλανδία υπόβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης του χελιού, σύμφωνα με το άρθρο 5.1 του κανονισμού 1100-2007. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εφαρμόζει τις, τα μέτρα τα οποία είχαν προτείνει οι επιστήμονες, οι εμπειρογνώμονες προκειμένου να ανακτηθούν τα αποθέματα χελιού. Επομένως, τα μέτρα τα οποία έχει οθετήσει η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή όντως συνάδουν με τις απαιτήσει του κανονισμού του Συμβουλίου και όντω συμβάλλουν στην ανάκτηση των αποθεμάτων χελιού στην Ιρλανδία. Αν κατακλείδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο το οποίο το πρόγραμμα διαχείριση του χελιού που εφαρμόζει το Υπουργείο Επικοινωνιών Ενέργεια και Φυσικών Πόρων πληρούν τι προποθέσει που ορίζονται στον κανονισμό 1100-2007. Επίσης, θα πρέπει ε, να αναλαμβάνεται αυτή η ενδεδειγμένη δράση σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τοπικές και περιφερειακέ ιδιαιτερότητε. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι ο κανονισμός αυτός περιγράφει αποκλειστικά και μόνο τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί ή την ανασύσταση του αποθέματος, επιτρέποντας ποσοστό διαφυγή στη θάλασσα τουλάχιστον 40% των χελιών. Η απόφαση ως προς τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου επαφείται εξ ολοκλήρου στα κράτη-μέλη. Ω εκ τούτου εναπόκειται στα κράτη-μέλη να επιλέξουν τα μέσα για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου. Η Ιρλανδία επέλεξε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία αξιολόγησε το ISIS, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ασύσταση του αποθέματο χελιού. Επιπλέον, εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, η Ιρλανδία συμβουλεύτηκε παρκώς τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο έγκαιρη δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη το 2008. Ευχαριστώ. Κυρία Μάρκιν. Thank you, Madam Chairperson. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν ε, ανέγνωσα καλά την, την μισή διάταξη, δεν γνώριζα όμως το θέμα πρόκειται να φύγει σήμερα. η <clears throat> τελευταία δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ότι όντως η ε, επίτευξη του στόχου εναπόκειται στα κράτη-μέλη, αλλά ότι η Κομισιόν το δήλωσε ξεκάθαρο το θέμα, θα πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση για όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στον τομέα τη κοινή ελευθερικής πολιτικής και σύμφωνα με την αναφορά η διαβούλευση με τους άλλους έγινε με καθυστέρηση αφού δηλαδή είχαν ληφθεί οι αποφάσει και ω εκ τούτου δεν λήψαν υπόψη οι θέσει του. Αυτό που θα πρέπει να λέμε είναι να υπάρχουν διαβουλεύσεις μεν αλλά να εισακούονται και οι ενδιαφερόμενοι διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη λοιπόν οι θέσει των διαφορεμένων. Και το λόγο που το λέω αυτό είναι διότι όταν οι Ιρλανδικέ αρχέ ήταν σε θέση να λάβουν την εν λόγω απόφαση, εάν δούμε όμω ότι ο ΦΑΣ που ελήφθησαν στην Βόρεια Ιρλανδία που βρίσκονται ακριβώ στα σύνορά μα στη Σκοτία και στη Γαλλία, που και θέσει είναι κοντινέ χώρε και ξέρουμε ότι τα αλλιεύματα ε, μετατοπίζονται, μετακινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη, καμία αυτέ αυτές τις ε, χώρες δεν ζήτησαν ε, να καταργηθεί απολύτως η αλία. Σε αυτή την περίπτωση ο Αλίας Χελιού πιστεύει πως στην περίπτωση των υπολείπων χωρών υπήρξε μία διαβούλευση ενώ στην Ιρλανδία αυτό δεν συνέβη διότι κάποιοι από τις απόψεις τους ε, δεν, λήφθηκε δεν υπόψη. Τώρα και έχω μια ερώτηση προς την Επιτροπή, διότι όπως είπα δεν έχω έρθει εδώ με κάποια τεκμηρίωση, κάποια έγραφα. Ε, αυτό φταίω εγώ. Λοιπόν, θα μπορούσα να είχα τις ημερομηνίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή οι Ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν το σχέδιο διαχείρισης του χελιού. δεν το έχω ενώπιον μου, ξέρω ότι υπήρχε μια προθεσμία τέλη Δεκεμβρίου του 2008. Ακριβή ημερομηνία δεν την έχω υπόψη μου, δεν την έχω μαζί μου, αλλά υπήρχε προθεσμία για τα Δεκέμβριο του 2008. Τώρα θυμάμαι. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα δεν έχω δώσει προφορίες, αλλά να τονίσω πως η διαβούλευση θα πρέπει να γίνεται και να λαμβάνονται υπόψη κάποιες από τις προτάσεις ε, σε που γίνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Καμία από τις προτάσεις που υπευρύθησαν λήφθηκε υπόψη και αναφέρομαι ότι σε άλλα κράτη τα οποία είτε συνορεύουν με την Ελλάδα είτε βρίσκονται πολύ κοντά οι απαντήσεις και οι θέσεις ε, των ε, ενώσεων των αλλιέων ελήφθησαν υπόψη. Μόνο στην ε, δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν ελήφθησαν υπόψη και υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Δεν βλέπω λοιπόν πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια τέτοια απαγόρευση. Έχω την αίσθηση ότι τίθεται ένα πολύ γενικότερο ζήτημα με την παρέμβασή σα αυτή ε, αν λάβουμε υπόψη ότι φαίνεται πως τα μέτρα που έχει λάβει η Ιρλανδική κυβέρνηση είναι αποτελεσματικά, είναι υπέρ της, ε, ε, είναι κατά της μείωσης του χελιού, αλλά απλώς υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν τα έχουν εφαρμόσει. Επομένω, το ζήτημα δεν έχει σχέση άμεση μόνο με την συμμετοχή των αλλιέων στην, στο συγκεκριμένο ψήφισμα, στη συγκεκριμένη οδηγία, αλλά και με το πόσο αυτή η οδηγία έχει ισχύ και για τις άλλες χώρες Ευρώπης. Αυτό είναι ένα άλλο ε, πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα έπρεπε ίσως να το δούμε δεν ξέρω αν υπάρχει να το δούμε εμείς ως Επιτροπή ή κάποιος άλλος. Η πρόταση είναι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την request opinion from Fisheries Committee. Ναι, αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε να καλέσουμε ε, να ζητήσουμε τη γνώμη και από την Επιτροπή Αλίας ε, σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι καλή ιδέα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Ναι, Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την ε, αποτελεσματική αντιπροεδρό μας. Περνάμε στο σημείο 15, αναφορά του Μάρτιν Κέριν, ο κύριος Γκονζάλες από την Κομισιόν. Έχετε λόγο. Όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου ζητήθηκε να σχολιάσω μία αναφορά που αφορά την αλία του Σολομού στην Ιρλανδία. Η αναφορά είναι του κύριου Μάρτιν Κέριν, Ιρλανδίου, ο κύριος Κέριν παραπονιέται ή μάλλον διαφωνεί με την πρόσφατη απαγόρευση της αλίας Σολομού με παρασυρώμενα απλάδια στην Ιρλανδία. Πέραν του ότι υπάρχει πληθώρα Σολομού, Είχαν αρχικά προβλεφθεί κάποιοι περιορισμοί στις ποσοστώσεις που είχαν υπολογιστεί σύμφωνα με κάποιες ε, επιστημονικές μελέτες και τελικά κατέληξαν στο να απαγορεύσουν απόλυτα, εντελώς δηλαδή, την ε, αλία με παραστρώμενα πλάδια. Ο κύριος Κέριν αναφέρει ότι τα αποθέματα Σολομού επηρεάζονται ιδιαίτερα από της, ε, από την εκτροφή Σολομού, κάτι το οποίο οδηγεί στην ανάπτυξη ενός μικροβίου, το οποίο επηρεάζει όμως και τους ε, Σολομούς ε, που ζουν ελεύθεροι. Αναφέρεται ο κ. Κέρνιον, δεν υπάρχουν ελλακτικές δυνατότητες και ό,τι δοκιμάστηκε μέχρι τώρα δεν ήταν αποτελεσματικό. Ο κύριος Κέριν θεωρεί πως θα έπρεπε να αναλάβει τη διαχείριση των αλλιευμάτων η ίδια η Ιρλανδία. Δηλαδή στην ε, η βιομηχανία της Ιρλανδίας, κάτι το οποίο σημαίνει λοιπόν οι Ιρλανδικές αρχές δεν είναι για αυτή τη διαχείριση του Σολομού. Τέλος, σχολιάζει πως η κοινή ελευθερική πολιτική δημιουργεί μια διακριτική μεταχείριση των Ιρλανδών αλλιέων, διότι οι ποσοστώσεις που τους χορηγούνται είναι πολύ κατώτερες από τις ποσοστώσεις που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ένωση. Η Κομισιόν μπορεί να κατανοήσει ότι τα παρασύρματα πλάδια δεν είναι η μοναδική απειλή για του πληθυσμού Σολομού. Αλλά αναγνωρίζω ότι η απειλή αυτή είναι σημαντική και πως οι Ιρλανδικέ αρχέ θα έπρεπε κάτι να κάνουν για να περιορίσουν, να απαγορεύσουν αυτά τα, τη χρήση αυτών των δικτυών. διότι με αυτόν τον τρόπο αλίας ε, εχμαλούζεται ακρίτως Σολομή στέλνοντας με κίνδυνο κατά αυτόν τον τρόπο τα αποθέματα του Σολομού βρίσκονται εκτό ασφαλών βιολογικών ορίων, συμπαραλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται σε ποταμού εκτό Ιρλανδία. Επαναλαμβάνω πως οι Ιρλανδικές αρχές ήταν υποχρεωμένες να λάβουν αυτά τα μέτρα για την απαγόρευση Προτού να συμβεί κάτι τέτοιο, η Κομισιόν είχε εκφράσει ανησυχία τη και είχε ζητήσει να γίνουν μελέτε στην Ιρλανδία και την, ε, το, μεγάλο, το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτέ οι μελέτε συμπερίφθησαν σε ένα έγγραφο τη Κομισιόν όπου αναλύεται το συνολικό πρόβλημα που αφορά στην αλία Σολομού με παρασυρώμενα πλάδια και όπου καταλήγει λέγοντα ότι η επίλυση του προβλήματο θα πρέπει να δοθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος, διότι αυτή η αλία γίνεται στα χωρικά ύδατα των κρατών, ως εκ τούτου οι Ιρλανδικές αρχές ε, είναι σε θέση να λάβουν την κατάλληλη απόφαση. Όταν η Κομισιόν ενημερώθηκε ότι απαγορεύτηκε αυτή η αλία με τα παρασυρώμενα πλάδια. Εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για το ότι η Ιρλανδία έλαβε μια τόσο αποφασιστική και αποτελεσματική στάση. Αλλά αναφέρθηκε ότι υπήρχαν ε, ελάχιστες εναλλακτικές δυνατότητες ε, Εάν όμως ε, δεν απαγορευόταν η ε, αλία με τα παραστρώμενα πλάδια, τότε θα θέταμε σε κίνδυνο τα όλα, το όλο απόθεμα των, ε, του Σολομού. Φυσικά, όπως ξέρουμε, τα, σε πολλές περιπτώσεις τα αποθέματα έχουν μειωθεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα διαφορετικό και όχι συγκυριακό. Τα μέτρα λοιπόν, είναι πρόβλημα διαφορετικό, θα έπρεπε να είναι και διαφορετικά. Και τα μέτρα που έλαβε η Ιρλανδία ήταν διαφορετικού χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διακριτική μεταχείριση της Ιρλανδίας ε, σε επίπεδο αληθικής πολιτικής, η Κομισιόν πιστεύει ότι, μάλλον ε, ξέρει ότι όταν ε, <clears throat> ότι μετά από την εισαγωγή της ε, κοινής λήψης πολιτικής τα ένομα συμφέροντα της Ιρλανδίας ελήφθησαν πλήρως υπόψη στις λεγόμενες προτιμήσεις της Χάγης. Και η Ιρλανδία είχε το δικαίωμα να αναπτύξει την, τον αλληλευτικό της κλάδο όπως προβλεπόταν ήδη μέχρι και η Ιρλανδία διατήρησε αυτό το δικαίωμα και οι προτιμήσεις της Χάγης όπως ονομάστηκαν διατηρήθηκαν <clears throat> κατά τη δικασία της κατανομής αλληλευτικών δυνατοτήτων και κάθε Δεκέμβρη που αποφασίζονται οι πιστοστός για την επόμενη χρονιά τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται στην Ιρλανδία σύμφωνα με το πλαίσιο των προτιμήσεων της Χάγης. Και τέλος, για την ανάθεση της ε, διαχείρισης ε, των αλευτικών αποθεμάτων από την ίδια την Ιρλανδία, τόσο, τόσο ο Σολομός όσο και τα καβούρια, αυτά είναι ζήτημα που άπτονται της ε, Ιρλανδικής αρμοδιότητας Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και ένα ζήτημα συνθήκων, διότι η Αλία εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο απάντησα στο, την αναφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Συμφωνώ με συγγνώμη. με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αλία με παρεσυρώμενα δίχτυα, την αλία Σολομού. Για τα υπόλοιπα ζητήματα θεωρώ ότι δεν εμπίπνουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας και θεωρώ ότι μέσω της αναθεώρησης κοινή ελευτικής πολιτικής θα διευθετηθούν τα προβλήματα αυτά και όπως ξέρετε την αναθεώρηση αυτή έχει σχεδόν ξεκινήσει. Συμφωνώ και εγώ. Στο σημείο αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε πως ε, μπορεί να κλείσει η εν λόγω αναφορά. Περνάμε στο σημείο 16. Για την τα μεταβίβαση πρέπει να δει τη χορήγηση ανάπτυξη στην Ιρλανδία. Αναφορά του Τόμας Ντόρνη και στην επόμενη του Τόμα Σουάρκ για την εφαρμογή της αλλογορήτρας ε, είναι παρόν ε, ο αναφέρον κύριο Τόμας Ντόρνη που δίνει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Η αναφορά μου έχει να κάνει με το ότι όταν μέλη της οικογένειάς μου κάνουν μια αίτηση κατασκευής στο δικό μας ουσιαστικά χώρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια αίτηση, η χορήγηση αυτή άδεια καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Θεωρώ ότι η περίοδος που είχε καθοριστεί είναι ιδιαίτερα άδικη, ότι είναι ιδιαίτερα μακροχρόνια. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά κριτήρια, τα οποία όμως θα πρέπει να συνδέονται περισσότερα περισσότερο με τις ιδιαιτερότητες περιοχής και επίσης δίδονται πάρα πολλοί περιορισμοί όσον αφορά την ε, συγγένεια που έχει κανείς με το άτομο το οποίο κατέχει την περιοχή, που έχει την της περιοχής και ε, προβλέπεται μια πάρα πολύ αυστηρή διαδικασία για την υποβολή της άδειας οικιστικής ε, ανάπτυξης και για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντηση που δόθηκε μας λέει ότι έχει ε, ζητήσει από τον Ιούνιο 2007 τις αρμόδιες αρχές να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να δει αν τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται για την χορήγηση άδεια όντω βασίζονται στα σωστά κριτήρια και αν συνάδουν τα κριτήρια αυτά με τα άρθρα 43 και 56 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα, οι συνθήκες αυτές για τη χορήγηση άδειας οικιστικής ανάπτυξης υφίστανται ακόμα στο Galloway της Ιρλανδίας και θεωρώ ότι Πρέπει να γίνει ακόμη μια διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στοιχεία που τη έχουν δοθεί από την Ιρλανδία δεν αρκούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και τώρα περνάμε στην επόμενη αναφορά, ο κ. Τόμα Σακίνη. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ονομάζομαι Τόμας Σάρκη, είμαι και εγώ από την Ιρλανδία, το Candy Line. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή σας να διατηρήσει την αφορά μου ανοιχτή και θα ήθελα να δοθούν και περισσότερες πληροφορίες. Η περίληψη της αναφοράς μου δεν αναφέρεται στο πιο σημαντικό τμήμα της αναφοράς μου που έχει να κάνει με την πρόσβαση, την ίση πρόσβαση στην ε, αγορά ε, ιδιοκτησίας και στη χρησιμοποίηση της ρήτρας περί προβλέπεται από την Ιρλανδική νομοθεσία προηγούμενη συμφωνία ανάμεσα στην, στον Ετούντα και την αρχή που χορηγεί την άδεια. Πρέπει να προβλέπεται λοιπόν η συμφωνία αυτή, η οποία είναι γνωστή και ως ρήτρα, ρήτρα περί χρήση κτησίας, που προβλέπεται για μια περίοδο συγκεκριμένοι 5-7 ετών και μεγαλύτεροι. Δεν είναι όμως αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Οι κατευθύνσει γραμμέ που χρησιμοποιούνται στην Ιρλανδία από το 2005 και μετά επιβάλλουν ρήτρα περί ε, χρησικτησίας που δημιουργούν ε, περαιτέρω γραφειοκρατία που τελικά επιβαρύνει αυτή τα άτομα που είναι ιδιοκτήτες συγκεκριμένων κατοικιών. Το πρόβλημα λοιπόν το δικό μου είναι ότι ε, οι κατευθύνες γραμμές περί χωροταξίας του 2005 δίνουν δυνατότητα opt-out εξαίρεσης για κάποιες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που τελικά πρημοδοτούνται από το σύστημα αυτό. Αντίθετα βρίσκονται σε πάρα πολύ δεινή θέση οι ίδιοι οι ιδιώτες, οι διοκτήτες πάρα πολλές φορές, που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα της κρίσης και πολλές φορές επιλέγουν να πουλήσουν την κατοικία τους προκειμένου να καταφέρουν να αποκτήσουν περισσότερους πόρους. Στην προσπάθειά τους να κάνουν κάτι τέτοιο, έρχονται αντιμέτωποι με την Ιρλανδική νομοθεσία που αυτή τη στιγμή θέτει εμπόδια στην πώληση αυτή. Από την άλλη βλέπουμε όταν υπάρχει μια τράπεζα ή ένας χρηματοπιστωτικός ε, οργανισμός ο οποίος αγοράσει την ιδιοκτησία αυτή, τότε τα εμπόδια αυτά τα οποία θέτει η ενας χρηματοπιστωτικος οργανισμος ο οποιος αγορασει την διοκτησια αυτη τοτε νομοθεσία δεν εφίστανται πλέον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μία τράπεζα, ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να πουλήσει ένα κτήμα ή ε, ένα σπίτι σε οποιονδήποτε άλλον αγοραστή, πιθανό αγοραστή στον κόσμο, ενώ ο ιδιώτης, ο ιδιοκτήτης του α, κτήματος ή του σπιτιού επιτρέπεται να το πουλήσει μόνο σε, κάποιον ο οποίος θα κατοικεί σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ακτίνα. Ε, ο εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ. Θα απαντήσω στους δύο αναφέροντες σε ό,τι αφορά ε, της τρίτρα μεταβίβασης. Σε ό,τι φορά την άλλη αναφορά θα απαντήσει ο συναδελφός μου. Τώρα θα ήθελα να κάνω διαφοροποίηση δύο ζητημάτων. ή αναφορές αφορούσαν την αμεροληψία της μεταβίβασης που ε, υποχρεώνει τους αγοραστές ε, να κατοικούν στο οικία για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να αναφέρω πως ε, η Κομισιόν δεν μπορεί να δράσει παρά μόνο σε θέματα που αφορούν διακριτική μεταχείριση στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας είτε των κεφαλαίων είτε των προσώπων, ελευθερία εγκατάσταση κλπ. Όπως ε, αναφέρθηκε στις απαντήσεις, η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάση στην Ιρλανδία εδώ και δύο χρόνια, διότι εξετάζοντας ε, μία σειρά ε, προγραμμα... αναπτυξιακών περιφερειακών προγραμμάτων, παρατηρήσαμε ότι κάποιες, κάποιοι όροι για την κατασκευή κατοικιών στην στην επαρχία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως διακριτικοί όροι. Όπως παραδείγματο χάρη η ανάγκη να κατοικεί κανείς ήδη στην περιοχή για να λάβει την άδεια οικοδόμησης ή να κατοικεί η οικογένειά του, οικογενειακά πρόσωπα κλπ. Συγγενικά. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που είναι αδύνατο να προωθούν από Ευρωπαίους κατοίκους άλλων κρατών μελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ρήτρα για την εκ των υστέρων κατοίκηση, βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι αποτελεί διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με περιορισμούς πρόσβαση στην στέγη, δηλαδή ο νόμος Ράις του 2002, όπου το δικαστήριο διευκρίνησε ότι τα κράτη-μέλη μπορούσαν να επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς σε ό,τι φορά την ε, εγκατάσταση για ελευθερεύουσα οικία, κατοικία για να υπάρξει μια οικιστική πολεμική ρύθμιση. μέσα από το πλαίσιο λοιπόν αυτού των περιορισμών αναφέρει η νομολογία του δικαστηρίου θα πρέπει να θέσουμε και τις ε, δυνατότητες της Κομισιόν. Τα κρατημέλη μπορούν να επιβάλλουν κάποιες ε, διατάξεις ε, για θέματα πόλεοδομίας, οικιστικής ανάπτυξης κλπ. εάν κρίνουν πως ορισμένες περιοχές, ορισμένα τμήματα της επικράτειας θα πρέπει να τύχουν περιορισμένης ανάπτυξης. Εδώ μιλάμε για όλες τις ρήτρε ε, που προανέφερα, μιλάμε λοιπόν και για ανάπτυξη σε περιοχές υπαίθρου. Δεν μιλάμε για πωλήσει κατοικιών ε, σε αστικές περιοχές. Λοιπόν, στις συζητήσεις που είχε η Κομισιόν με τις Ιρλανδικές Αρχές, οι ρήτρε μεταβίβασης θεωρήσαμε ότι ήταν ε, πιο ισότιμες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ε, σε, μια, σε, σε κάποια περιοχή της Ισλανδίας ε, όπως αναφέρει και η απόφαση του δικαστήριου. Φυσικά αυτοί οι περιορισμοί θα πρέπει να παραμείνουν περιορισμένοι και αφορούσαν συγκεκριμένες γεωγραφικές ε, περιφέρειες. Θα μπορούσε η κατάσταση να εξεταστεί από διαφορετική οπτική γωνία εάν είχαν επιβληθεί παρόμοιες ρήτρε ε, σε όλη την επικράτεια, σε χωριά, πόλεις κλπ. Αλλά αυτές οι ρήτρε δεν αφορούν παρά μόνο την Ήπεθρο και ε, και τα όσα αναφέρονται περί διακριτικής μεταχείρισης ε, αποτέλεσαν αντικείμενο αίτηση τροποποίησης προς το αρμόδιο Υπουργείο της Ιρλανδίας, το οποίο ζήτησε από τις περιοχές να εξετάσουν τα οικιστικά αναπτυξιακά προγράμματα για να δουν πως ε, τέτοιες ε, προϋποθέσεις εφαρμόζονται, υλοποιούνται και να μην συνεχίσουν τις εφαρμόζουν σε περίπτωση εγκατάστασης ε, ατόμου που επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή. Γνωρίζουμε πως ορισμένα περιφερειακά πολεμικά σχέδια πρόκειται να τροποποιηθούν και περιμένουν πριν πληροφορίες από τις ελληνικές Αρχές. Ό,τι φορά τώρα την ερώτηση που έθεσε ο κ. Σαρκέ, η μνήα στο ότι σε περίπτωση δυσκολιών ε, αποπληρωμής ή πώλησης ε, ιδιοκτησίας από τράπεζα. Το πρόβλημα είναι το αυτό. Θα πρέπει να βρούμε την επιβολή διάκρισης έναντι σε πολίτες ε, άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Αυτή η ρήτρα αποτελεί διακριτική μεταχείριση Ευρωπαίων πολιτών που θα επιθυμούσαν να εγκατασταθούν ενδεχομένω στην Ιρλανδία. Κατανοώ το πρόβλημα που, ε, που θίγεται μάλλον με αυτήν την ανισότητα που μπορεί να προκύψει, αλλά βρισκόμαστε στο πλαίσιο μιας διακριτικής μεταχείρισης που μπορούσε να καταπολεμηθεί με την ε, ρύθμιση περί, του, περί εγκατάστασης. Χάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο τελευταίο της σχόλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αφορά του κύριου Σάρκη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σαφής, είπε ότι ως ιδιώτης δεν μπορεί να πουλήσει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να πουλήσει σε έναν Έλληνα, σε έναν Βρετανό, σε έναν Γερμανό. Το επιτρέπεται να πουλήσει μόνο σε κάποιον ο οποίος ζει μια συγκεκριμένη απόσταση από το σπίτι του. Κοντά ουσιαστικά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν μπορεί να πουλήσει κανείς ένα σπίτι, τότε ο Γερμανός, ο Έλληνας, ο Βρετανός πολίτης δεν μπορεί να αγοράσει αντίστοιχα ένα σπίτι στην Ιρλανδία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν είναι απόλυτα πεπισμένη ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ελευθερία τη εγκατάσταση. Σίγουρα όμω, θα πρέπει να δερβηνηθεί ακόμα περισσότερο το ζήτημα αν μη τι άλλο και αυτό ακριβώ ζητά και ο αναφέρον. Και νομίζω ότι υποστηρίζει πολύ καλά το πρόβλημά του αυτό και όντω και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματο. Τώρα, το άλλο ζήτημα το οποίο συνδέεται βέβαια με το πρώτο είναι ότι σε μια πρώτη φάση, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τι Ισλανδικέ Αρχές, είπαν ότι υπήρχαν διάφορα ζητήματα, τα οποία ενδεχομένω να μην συνάδουν με το 43 και 56, τα άρθρα 43 και 56 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μάρτιο του 2009, ε, το ίμιση των περιφερειών τελικά είπαν ότι τα σχέδιά του συνάδουν με το περιεχόμενο της εγκυκλίου. Θα ήθελα να γνωρίσω τι έγινε με το υπόλοιπο ήμιση, e δηλαδή αν πρέπει όντω να συμμορφωθούν με την εγκύκλιο. Τότε όλε οι περιφέρειε θα πρέπει να συμμορφωθούν, έτσι δεν είναι. Και ειδικότερα επειδή ο κύριο Ντούρι είναι από το Galway τη Ιρλανδία, θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν η περιφέρεια αυτή έδωσε μια απάντηση όσον αφορά το περιεχόμενο της εγκυκλίου, την μπροστά μου θα είμαι και πολύ σύντομη, ξέρω ότι περνάει ο χρόνος. Έχω πάντως μπροστά μου ένα αντίγραφο του σχεδίου ε, ανάπτυξης για αυτή την ε, περιφέρεια, όπου αναφερόμαστε σε περιορισμένη δυνατότητα οικοδόμησης για συγκεκριμένες οικογένειες και ότι ε, θα μπορούσε να δοθεί μόνο άδεια σε θυγατέρες και ιούς στην, στο αγρόκτημα των γονέων τους θεωρώ ότι η διάταξη αυτή ακόμα περιέχει την ρήτρα αυτή τη διακριτική, της διακριτικής μεταχείρισης την οποία εξετάζει, εξέταζε τουλάχιστον στην αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αναφερόμαστε εδώ πέρα στο σχέδιο ανάπτυξη 2009-2015. Δηλαδή η ρήτρα αυτή θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετά εκρεμή ζητήματα ακόμα και μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να τα επεξεργάζεται, δεν νομίζω ότι έχουν αποσαφινιστεί. Και ένα τελικό ερώτημα που έχω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να μου δοθεί και μια γραπτή απάντηση, γιατί δεν θα ήθελα να καταναλώσω τον χρόνο της συνεδρίασής μας, από ό,τι καταλαβαίνω, ενδεχομένως να έχουν υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις αστικές περιοχές, όσον αφορά την διακριτική μεταχείριση. Έχει συμβεί τελικά κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερα για το ζήτημα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα και για τις δύο αναφορές και για την πρώτη να παραμείνουν ανοιχτέ γιατί χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you very much. I too... Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το τελευταίο σημείο που ανέφερε η Κομισιόν απαντώντας στην αναφορά του κ. Δηλαδή κάποια ανομαλία που φαίνεται ότι υπάρχει. Όταν ένα μεμονωμένο άτομο, μια οικογένεια μπορεί να πουλήσει το σπίτι μόνο στην περιοχή, σε άτομα της περιοχής και όχι από παντού. Άρα, εάν κάποιος βρίσκεται σε, σε οικονομικές δυσκολίες και ανακτά η τράπεζα το, το ίδιο το σπίτι αυτό, μπορεί να το πουλήσει όποιον θέλει και να πετύχει βέβαια πολύ ψηλότερη τιμή παρά αυτό το άτομο το οποίο μπορεί να πουλήσει μόνο στους γείτονες. Θα ήταν καλό νομίζω να έχουμε μια διευκρίνηση από τις ελληνικές αρχές αυτού του σημείου, Πρόεδρε. Darei prima la parola. Ah, prego, Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Αλλά έχουμε τόσες συνεδριάσεις, στις οποίες θα πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα παρόντες. Ο λόγος που ήρθε ως αναπληρωτής της Επιτροπής Αναφορών είναι ακριβώς να υποστηρίξω αυτές τις ε, αναφορές. Μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Ρίγαν και την κυρία Τεπρούν να μην είναι ανοιχτή η αναφορά αυτή. Για κάποιους λόγους υπάρχουν πολλοί περίεργη περιορισμή στην Ιρλανδία όσον αφορά το θέμα των ε, πολυδομικών προγραμμάτων. Και αυτό που εξετάζουμε εδώ στις περισσότερες περιπτώσει είναι αγροτικά σπίτια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιρλανδία είναι μια αγροτική κοινωνία. Και εδώ και πολλά χρόνια οι διατάξεις εκεί γίνονται όσο πάει και πιο αυστηρές. Και φαίνεται η απόφαση είναι να σπάψει να είναι αγροτική η κοινωνία της Ιρλανδίας και να την μετατρέψουν οι αρχές σε μια αστική κοινωνία. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον να αφήσουμε ανοιχτή την αφορά για να ακούσουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει τις τρεις ε, αναφορές. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Μισελ. Α, όχι, συγγνώμη. Στον εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ. Είμαι εδώ για την αναφορά του κ. Μπέβη αλλά γενικά όσον αφορά την ε, Ιρλανδική πολυδομική νομοθεσία και ε, υποτιθέμενες διακρίσεις που παρεμποδίζουν τους ε, νεοφερμένους να κατασκευάσουν σπίτι κατοικίες. Η δική μου η αναφορά στην οποία είμαι αφορά έναν Ολλανδό πολίτη, όπου εδώ αναφέρομαστε σε μια δυνατότητα διάκρισης όσον αφορά την ε, θεγημερία του. Και λέμε ότι αποσρίφηκε η αίτηση τη γυναίκας του για μια κατασκευή, γιατί υποτίθεται ότι δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει πραγματικά ανάγκη εγκατάστασης. Αυτό σχετίζεται και με την διαδικασία που παραβάσει κατά της Ιρλανδίας του 2007. Κατόπιν συζητήσεων με την Κομισιόν, οι Ιρλανδικές αρχές το Σεπτέμβριο 2008 έστειλαν μια εγκύκλωση σε όλες τις Ιρλανδικές περιφέρειες ε, ζητώντας να εξασφαλίσουν ότι είναι ε, οι διατάξεις που εφαρμόζουν ευθυγραμμισμένες με την κοινοτική νομοθεσία οι μισές περιφερειές δήλωσαν ότι είναι συμβατές. Ε, οι άλλες είπαν ότι τροποποιούν αυτές τις στιγμές την ε, τους, ε, το πολεμικό τους προγραμματισμό για να μπορέσουν να ευθυγραμμιστούν με την κοινωτική νομοθεσία. Όσον αφορά τις απαιτήσει του κοινοτικού νόμου, θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι οι περιορισμοί για κατασκευές στην Ήπεθρο δεν είναι απαραίτητα ασύμβατες προς τον νόμο της Ένωσης. Μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί εφόσον εφαρμόζονται κατά μη διακριτικό τρόπο. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να ζητήσω από τη συνάδελφο να διευκρινίσει. Euh, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην πρώτη μου απάντηση έκανα ξεκάθαρα μια διάκριση μεταξύ των όρων εγκατάστασης μετά την αγορά και των όρων πριν από την αγορά ή πριν από τη χορήγηση οικοδομικής άδειας. όσον αφορά τη δυνατότητα οι τράπεζες να ξαναπολύσουν την ε, ιδιοκτησία αυτή σε περίπτωση οικονομικών δυσκολιών του ιδιοκτήτη σε πιο ευρύ ε, κοινό. Ενώ ο ιδιοκτήτης θα μπορούσε να πωλήσει μόνο σε αυτούς που είναι εγκαταστημένοι ήδη στην περιοχή. Αυτό είναι μια διάκριση. Είναι παράβαση. Εάν όμως υπάρχει μια διάταξη που να λέει ότι ο καινούριος ιδιοκτήτης πρέπει να κατοικήσει τουλάχιστον 5 ή 10 χρόνια την κατοικία αυτή που αγόρασε, εκεί είναι πιο δύσκολο να αποδειχθεί μια διάκριση, γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που έρχονται ε, να εγκατασταθούν για να εργαστούν στην Ιρλανδία πρέπει να αποδείξουν ότι κατοικούν. Υπάρχουν ε, κάπου 30 κομιτείες στην Ελλανδία. Οι μισές, όπως σας είπα, απάντησαν στην Κομισιόν ότι είναι σύμφωνες με την νέα οδηγία. Οι άλλες μισές αυτή τη στιγμή τροποποιούν τις διατάξεις τους. Καμιά φορά υπάρχουν περιφερειακά σχέδια που λήγουν. Και όλα αυτά τα σχέδια αναθεωρούνται. Και μιλάμε εδώ για έγγραφα εκατοντάδων σελίδων, γιατί καλύπτουν όλες τις πτυχές ε, τοπικής, ε, αγροτικής ε, και πολυοδομικής ανάπτυξης. Δεν έχουμε λοιπόν ακόμα τελικά στοιχεία. Ελπίζουμε σύντομα να τα λάβουμε και κάναμε τη σχετική έκκληση στις Ισλανδικές αρχές. Ελπίζω να απάντησα στις ε, ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ζητήσω από την εκπρόσωπο της Κομισιόν εδώ, στην περίπτωση που η σχέση ανάμεσα το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η ηθαγένεια είναι πολύ στενά συνδεδεμένες και αυτό δεν παραβιάζει κάποια βασική διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι ακόμα. Έχουν υπάρξει προηγούμενοι, υπάρχουν και άλλες χώρες όπου έχουμε παρόμοιους, παρόμοιες ρυθμίσεις και τρίτον τα 12 κράτη-μέλη που προσφάτως εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν παρόμοιες ρήτρε που αφορούν το θέμα της ε, ιδιοκτησίας διότι εάν ε, ούτως έχει το πράγμα να σας πω ότι Παρακαλείτε ο μιλής να μιλάει στο μικρόφωνο ότι κάτι παρόμοιο εάν ε, και εφόσον υπάρξει δημιουργεί έκπληξη τόσο σε δικαστικούς ε, χώρους όσο και στους πολιτικούς και φαντάζομαι και ποια θα είναι η αντίδραση των Ευρωπαίων της Δύσης ε, όταν σε κάποια αυτές τις χώρες θα μπορούσε καν να θίξει, να αναφέρει δηλαδή παρόμοιες ρήτρε που ισχύουν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εάν κατάλαβα σωστά, ένα από του εκπρόσωπου της Κομισιόν είπε ότι αν υπάρχουν ε, καλοί ε, λόγοι, δικαιολογημένοι λόγοι για του περιορισμού αυτούς, μπορούν να παραμείνουν. Θα ρωτήσω στον Κομισιόν, έχουν κατευθυντήριε γραμμές για κάτι τέτοιο, έχουν κατάλογο των περιορισμών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποδεχθεί. Και δεύτερον, ποια είναι η άποψη Κομισιόν σε τομεί στο Γκέλταχ στην Ιρλανδία, όπου ομιλείται η Ιρλανδική γλώσσα, βρίσκεται όμως υπό τεράστια πίεση και οι τοπικές αρχές σε ορισμένες από τις περιοχές αυτές έχουν επιβάλει όρους γλωσσικούς, ότι θα πρέπει δηλαδή να μιλάνε την τοπική γλώσσα, τα Ιρλανδικά, αυτοί που εγκαθίσταν εκεί. Αυτό είναι σύμφωνο με αυτό που η Κομισιόν θεωρεί την, ε, την, ε, το συμβατό με την συνθήκη. Very briefly, two questions for the Commission. Πολύ σύντομα δύο ερωτήσει για την Κομισιόν μετά από αυτά που μας είπαν αναφέρθηκαν στο ότι εάν η τράπεζα πουλήσει το σπίτι αυτό, τότε αυτή η ρήτρα εγκατάσταση θα ισχύει και για τον Έλληνα, τον Βρετανό κλπ. Κατάλαβα τι είπαν, αλλά δεν ασχολούνται όμως με το θέμα ότι αν οι ιδιοκτήτες, οι οικογένειες θέλουν να πουλήσουν δεν μπορούν να πουλήσουν σε έναν Έλληνα, Γερμανό ή Βρετανό. Επιτρέπεται να πουλήσουν μόνο σε κάποιον που είναι γείτονας ήδη. Αυτό σημαίνει ότι ένας Γερμανός, Πολωνός, ε, Βρετανός, Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει αυτό το σπίτι. Και πιστεύω ότι αυτό είναι μια διάκριση που βασίζεται στην ηθαγένεια ή στην υπηκότητα όπως ε, πρότεινε και ο συνάδελφος. Άλλη ερώτηση που θέλω να υποβάλω προς την Κομισιόν μας είπε ότι έλαβαν απαντήσεις από τις μισές εν λόγω περιφέρειας. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι απαντήσεις που πήραν είναι ικανοποιητικές. και ότι δεν τίθεται θέμα ότι αυτές οι απαντάσεις δεν είναι συμβατές με τα άρθρα 43 και 56 συνθήκης. Να δώσω το λόγο στον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν για να απαντήσει τις ερωτήσεις, αν και εν μέρει νομίζω πως έχουν απαντηθεί στην ανακοίνωση που έχει γίνει από δύο δήμα από την Κομισιόν ως απάντηση και στην ανακοίνωση που έκανε η Κομισιόν ότι υπάρχει λοιπόν πρόθεση να παρακολουθήσουν εκ του εξελίξεις για να δουν κατά πόσον υπάρχει παράβαση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερής κυκλοφορίας προσώπων. Αν υπάρχουν λοιπόν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις να δοθούν τώρα, αλλά σύντομα παρακαλώ, διότι έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά όρια. Ναι. Με συγχωρείτε. Sì, però dopo do la, la, la replica ai firmatari. Εντάξει, θα λάβετε μετά το λόγο, αφού απαντήσει η Κομισιόν. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω σε ερωτήσει. Η πρώτη που αφορά το σχετισμό μεταξύ διοκτησία και υπηκότητα. Το άρθρο 12 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει διακρίσεις βάσει της μέσα στα πλαίσια της εμβέλειας της συνθήκης. Και βέβαια το θέμα της εγκατάστασης της οικοδόμησης ε, οικίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή της ε, συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και καμία διάκριση. Αλλά Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν τα πάντα μέσα στην ευέλεια της συνθήκης και ότι δεν είναι τα πάντα απαραίτητο διακρίσεις. Παραδείγματο χάρη, καταστάσεις που δεν αφορούν διαμεθοριακά θέματα δεν εμπίπτουν στην ευέλεια της συνθήκης. Παραδείγματο χάρη, οι Ιρλανδοί υπήκοοι μέσα στην Ιρλανδία. η ελευθερία κίνηση τους μέσα στην Ιρλανδία κλπ. δεν υπάρχουν στη συνθήκη. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει διάκριση βασιζόμενη στην υπηκότητα. Από την άλλη μεριά στην ε, νομολογία της Ευρωπαϊκής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρεται ότι διαφορετική μεταχείριση δεν σημαίνει απαραίτητο διακρίσεις υπό το πνεύμα τη συνθηκη γιατί μπορεί να δικαιολογούνται. Και λέει ότι η διαφορά μεταχείριση θα πρέπει να είναι αναλογική και η αναλογικότητα αυτή εφαρμόζεται κατά περίπτωση. βάσει κάστοτε αξιολόγηση. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένε καταστάσεις στι οποίε το δικαστήριο λέει ότι αυτό είναι αποδεκτό. Άλλες φορές λέει ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η διακριτική μεταχείριση. Και όσον αφορά το θέμα της γλώσσας, που αναφέρθηκε, Καταρχήν, αυτό είναι μια διαφορετική μεταχείριση. που έχει αντικές επιπτώσεις στους ε, υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τους Ιρλανδούς που δεν μιλάνε την ελληνική. η Κομισιόν σε σχέση με παρόμοια ε, θέματα όσον αφορά την πρόσβαση στη κοινωνική κατοικία στο Βέλγιο, σε ορισμένε περιοχέ, όπου αυτό εξαρτάται παραδείγματο χάρη δυνατότητα να μιλάει κανένα φλαμαδικά. Η Κομισιόν έχει κατά νου ε, μια, κάποια δράση κατά του κράτους του Βελγίου. Πρόεδρος, να προσθέσω κάτι. Αναρωτιόμουν σε σχέση με τα σημαντικά θέματα που δείξαμε χάρη σε αυτές τις αναφορές. Ποια είναι η γνώμη της Κομισιόν ε, σχετικά με την θέση τη της συνθήκη Λισαβόνας που έχει περάσει και την διαδικασία του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία και τα θέματα τα οποία εξετάζουμε τώρα. Δηλαδή, πώς εντάσσονται λοιπόν όλα αυτά στο πλαίσιο των αρχών που καθορίζονται στην χάρτη των δικαιωμάτων που εμπεριέχεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω πως η τελευταία ερώτηση θα είναι πιο δύσκολο να απαντηθεί. Θα απαντήσω όμως σε κάτι άλλο το πρώτο ερώτημά σας, ε, κατά πόσον υπάρχουν άλλα κράτη που εφαρμόζουν παρόμοιους κανόνες. Η Κομισιόν ε, αντιδρά μετά από υποβολή διαμαρτυριών. Έχουμε λάβει διαμαρτυρίες ε, από πολλά κράτη-μέλη, αλλά είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε εάν στις 27 κράτη-μέλη υπάρχουν παρόμοιες ρυθμίσεις. Γνωρίζουμε περιπτώσεις ε, στο Βέλγιο που υπάρχει κάποια γλωσσική ιδιαιτερότητα. Μα αυτό αποτελεί και μια πρόσκληση σε εσάς ε, να κάνετε κάποιες έρευνες. Ε, μιλήσατε για εξαιρέσεις. Η Αυστρία με την ένταξή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε να διατηρήσει μια, ένα μεταβατικό καθεστώς και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έφτασαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να εφαρμόζονται αυτές οι εξαιρέσεις κλπ. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τις ιδιοκτησίες. Παλιά υπήρχε κάτι παρόμοιο. Όπως είπε και ο συνάδελφος, τώρα μια παρόμοια απαγόρευση είναι κάτι το που δεν περνάει καν από το μυαλό. Δεν μιλάμε για λόγους ηθαγένειας. Μιλάμε για έμεσες ε, διακρίσεις, όπως στην περίπτωση της Ιρλανδία, δηλαδή να κατοικείς μεγάλη περίοδο σε άλλο κράτος μέλος πριν να μπορείς να αποκτήσεις οικία. Αυτό αποτελεί διάκριση για όσους κατοικούν εκτός Ιρλανδίας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ελέγξουμε εδώ τη διάκριση. Το να υπάρχουν και ε, κάτοικοι που να ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον και αυτό αποτελεί διάκριση. Δεν είναι δυνατόν σε κράτος μέλος ε, να περιορίσει το δικαίωμα ιδιοκτησίας ε, βασιζόμενο στην ηθαγένεια. Δύο κράτη, τρία αν θέλετε, γνωρίζω όπου υπάρχουν παρόμοιε περιπτώσεις, αλλά δεν αφορούν ε, στο ε, ιδιοκτησία, απλά οφείλονται στην ιδιάζουσα κατάσταση που επικρατεί στο Βέλγιο από γλωσσική σκοπιά. οι Ευρωπαίοι, και οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιδρούν άμεσα σε αυτού του είδους ε, διακριτικής μεταχείρισης και Πρόσφατα διάβασα ότι περίπου 9 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών κατοικούν σε άλλο κράτος ε, μέλος από αυτό της ε, καταγωγής τους. Όλο και περισσότεροι μετακινούνται για 6 μήνες ή ένα έτος και παρόμοιες διαμαρτυρίες ε, λαμβάνουμε συχνά στην Κομισιόν όταν υπάρχουν περιορισμοί στο κάποια δικαιώματα, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, υπάρχει και το διασυνοριακό στοιχείο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί με τρόπο απλούστερο ειδικά σε ό,τι αφορά κάποιες ε, δραστηριότητες ε, και να συνεχίσω λέγοντας πως ε, εάν η Κομισιόν έχει κάποια, κάποιο κατάλογο για, αυτές, για αυτούς τους περιορισμούς. Κοιτάξτε, κατευθύνες γραμμές παίρνουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο κανόνας που ανέφερα προηγούμενα μας οδήγησε στο να κρίνουμε ότι υπάρχουν μια φορά επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος σκεφτούμε μια περιοχή όπου ο τουρισμός αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της οικονομικής ζωής. Αν υπάρξει πρόβλημα, ας φανταστούμε μια ευρύτερη ρήπανση της περιοχής, όλη η οικονομική δραστηριότητα που στηρίζεται στον τουρισμό πάει, πεθαίνει, εξαφανίζεται. Δεν μπορεί να επιβιώσει η περιοχή διότι δεν θα υπάρχουν πλέον τουρίστες. Και το δικαστήριο έθεσε σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο περιορισμών δέχθηκε αυτή την αιτιολόγηση, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλου περιορισμού, όχι μόνο σε θέμα ιδιοκτησία, αλλά σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα. Και εξετάζουμε πάντα αν υπάρχει κάποια επιτακτική ανάγκη και αν αυτοί οι περιορισμοί είναι οι κατάλληλοι προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητό στόχο. Φυσικά, ό,τι αφορά στο περιβάλλον θα μπορούσε να αποτελέσει μια ε, επιτακτική, επιτακτικό λόγο όταν λοιπόν τα κράτη-μέλη ε, καταρτίζουν τα ε, πολυδομικά σχέδια ή τα χωροταξικά φροντίζουν να περιορίσουν τις Περιβαλλοντικέ επιπτώσει ε, και η Κομισιόν λοιπόν σε την περίπτωση μπορεί να δεχθεί τα επιχειρήματα του κράτους ε, αλλά ε, υπό την έννοια ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι να εφαρμοστούν αλλά και είναι ικανοί για την επίτευξη του στόχου. Οι περιορισμοί μπορούν να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη σε κράτος μέλος αλλά κάθε είδους δραστηριότητα δεν μπορεί να απαγορεύεται. Λοιπόν, είναι αυτό κάτι το οποίο ζητάει να λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο. Η Κομισιόν φροντίζει να το εφαρμόζει. Τώρα, σε όλη φορά το γενικό συμφέρον, τα ζητήματα ε, χωροταξίας και πολεμίου και πρέπει να φροντίζουν να προστατεύσουν την οικονομική ζωή κλπ. Ευχαριστώ. Θέλει κανένας από τους αναφέροντα να λάβει το λόγο. Ένα σημείο που μου προξένησε εντύπωση είναι ότι εδώ ο κύριος δίπλα μου είπε κάτι πολύ σωστό. Είπε ότι ε, στο Κόρ και στο Γκάλουι φαίνεται ότι θέλουν τελικά να περάσουν από την ανάπτυξη της υπαίθρου περισσότερο στην ανάπτυξη των πόλων. Θέλουν ουσιαστικά να διαμορφώσουν τις περιφέρειες αυτές περισσότερο αστικές περιφέρειες. Εγώ νομίζω όμως ότι ε, το ζήτημα θα πρέπει να μείνει ανοιχτό, ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες. Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, ε, αυτό με ικανοποιεί, με καλύπτει να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Επιτροπή Αναφορών που έλαβε υπόψη της αναφορά μου καθώς και τις άλλες αναφορές. Έμαθα πολλά πράγματα ακούγοντας την κατάσταση σε, όπως την περιέγραψαν οι ευρωβουλευτές στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνοψίζοντας θα ήθελα να πω ότι όντως υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες κηρύσουν πτώχευση και πάρα πολλές τράπεζες οι οποίες πλουτίζουν πουλώντας τα σπίτια τους και θα ήθελα λοιπόν αυτό να ληφθεί δεόντω υπόψη. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας πολίτης από ένα άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να αγοράσει από μένα το σπίτι μου παρά μόνο και μόνο όταν η τράπεζα το αγοράσει από μένα, μόνο τότε μπορεί το σπίτι μου να πουληθεί μέσω της τράπεζας όμως μόνο πλέον στον άλλο πολίτη της ε, άλλης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μειώνται οι δυνατότητες πώληση από τον ιδιώτη, από τον κάτοχο του σπιτιού. Εγώ σας ευχαριστώ που υποβάλατε αυτές τις αναφορές. Τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ακούσαμε και ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις. Θα προχωρήσουμε λοιπόν προκειμένου να ρίξουμε άπλετο φως στις υποθέσεις αυτές. Θα ζητήσουμε περαιτέρω γραπτές πληροφορίες από την Κομισιόν και θα δούμε κατά πόσο θα χρειαστεί να συνεργαστούμε και με άλλες κοινοβουλευτικές τροπές όπως η ΛΥΜΠΑ κλπ. Προσβλέπουμε λοιπόν σε μια έγκαιρη απάντηση από την Κομισιόν. Περνάμε στην επόμενη αναφορά, υπάρχει 17 του κυρίου Ράμς Μπότομ αφορά στις διακρίσεις λόγω ηλικίας από πλευράς Κομισιόν η κυρία Κριστίν Χόνερ. Σας ευχαριστώ. Ο αναφέρον είναι 70 ετών και αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς τη λήψη ενυπόθηκου δανείου λόγω των περιορισμών ηλικία που τίθενται από ορισμένου δανειστέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που κυμαίνονται από τα 65 στα 80 έτη και αφορούν στο ανώτατο όριο ηλικία για την άρση υποθηκών. Ο Ναφέρον πιστεύει ότι η περιγραφή σε κατάσταση αποτελεί διάκριση λόγω ηλικία. Αμφισβητεί την αναγκαιότητα μια τέτοια διάκριση Δεδομένου ότι, εν αντίθεση με άλλε οικονομικέ υπηρεσίε όπω ασφάλεια ζωή, τον υπόθηκο περιστατικό στοιχείο είναι το ίδιο ανεξαρτήτω ηλικία. Αναρωτιέται λοιπόν ο αναφέρον αν το ζήτημα αυτό αποτελεί τμήμα τη κοινοτική νομοθεσία και τι θα μπορούσε να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισχύον νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή Κοινότητα απαγορεύει τι διακρίσει λόγω ηλικία στην Προσχώρηση της, για τη χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Λέγεται μάλιστα ότι οι χρηματοστοτικέ υπηρεσίε έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν, έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν την ηλικία ενό οφειλέτη. Επομένω, η ηλικία αποτελεί πολύ σημαντικό συντελεστή κινδύνου, γιατί επηρεάζει τι δυνατότητε του οφειλέτη να αποκληρώσει το δανειό του. Και αυτό συνδυασμό με κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπως το καθεστώς απασχόλησης του οφηλέτη ή το αν είναι παντρεμένος ε, ή όχι. Ο αναφέρον λέει εδώ πέρα δεν θα πρέπει η ηλικία να αποτελεί περιοριστικό συντελεστή. Σε αυτό όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά ότι οι ε, δανειστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως έσχατη λύση και το, την παράμετρο της ε, ηλικίας, καθότι συνδέεται με τον ε, κίνδυνο. Επίσης, οι δανειστές μπορούν μπορούν να δανείσουν χρησιμοποιώντας τις προϋποθέσεις που κρίνουν αυτοί τις πιο, ότι είναι οι πιο αναγκαίες. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με μια πρόταση πρόσβασης όλων των πολιτών σε διάφορα προϊόντα της αγοράς, όπως και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η πρόταση αυτή εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο και πάλι όμως εδώ πέρα τα εθνικά, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν αυτά θα χρησιμοποιούν τον, την ηλικία ως καθοριστικό παράγοντα για την ε, χορήγηση τέτοιων υπηρεσιών ή για την πώληση χρηματοπιστωτικών ε, προϊόντων ο συναδελφός μου θα μπορέσει στη συνέχεια να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, η χρησιμοποίηση του ορίου ηλικία μπορεί αυτό να δικαιολογηθεί από το, ότι, από το επιχείρημα ότι ο φιλέτης δεν θα καταφέρει να αποπληρώσει το δάνειο. Μπορεί όντως να θυμηθεί απάντηση, πάντως σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι η χρησιμοποίηση του ορίου ηλικία αποτελεί παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Ε, Επιθυμεί να λάβει το λόγο. Νομίζω πως η απάντηση ήταν ε, αναλυτική, εξαντλητική και κάλυψε όλες τις πτυχές. Ε. Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι ότι κλείνει στο σημείο αυτό η αναφορά. Περνάμε στην επόμενη αναφορά, υπαριθμό 18, Κύριο κ. Κένεθα Μαλτέζικη Σταγένεια, σχετικά με εικαζόμενε παραβιάσει από τι Μαλτέζικε Αρχέ Κοινοτική Νομοθεσία για την αναγνώριση ισοτιμία των προσόντων. Νιωστή περίπτωση. Η Αντζέλικα Κόμεν από πλευρά Κομισιόν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αναφορά του κυρίου Κένεθα Αμπέλ έχει να κάνει με την αναγνώριση της σωτημίας προσόντων. Την 1η Οκτωβρίου, στην προηγούμενη συνεδρίαση δηλαδή, συζητήθηκε το ζήτημα αυτό και θελήσαμε να μάθουμε αν οι μαλτέζικες αρχές εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την αναγνώριση των προσόντων, την ισοτιμία των προσόντων. Έγινε επίσης μια βίντεο conference στις 24 ε, Ιουνίου, ήταν παρόν ο αναφέρον και συζητήθηκε το ζήτημα αυτό και σε άλλες επαφές που υπήρχαν μεταξύ των Μαλτέζικων Αρχών και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ο Ευρωβουλευτής που ασχολείται με τον αναφορά αυτή πιστεύει ότι έχει διευθετηθεί το ζήτημα, αλλά ότι ε, έπρεπε να δοθούν ακόμα περισσότερα στοιχεία. Θα ήθελα να σα δώσω τα στοιχεία αυτά τα οποία μπορούν να βεβαιώσουν την απόφαση αυτή. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιο ο αναφέρον υπέβαλε προ την Επιτροπή ένα αντίγραφο τη επιστολή που το έστειλαν από το Μαλτέζικο Επιμελητήριο Μηχανικών, που είναι η αρμόδια αρχή η οποία μπορεί να αποφασίσει για την επαγγελματική του επάρκεια. Η επιστολή είναι της 12 Οκτωβρίου και καταδεικνύει ξεκάθαρα το τα προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχει ο αναφέρον και αιτιολογείται μάλιστα η στάση αυτή του ε, Επιμελητηρίου Μηχανικών της Μάλτας. Οι Μαλτέζικες αρχές ε, όχι μόνο λαμβάνουν απόφαση γραπτός, αλλά στις 18 Αυγούστου κάλεσαν τον ίδιο τον αναφέροντα και του δώσαν τη δυνατότητα να μιλήσει περισσότερο για τα επαγγελματικά του προσόντα, για την επαγγελματική του εμπειρία, την οποία κατάφερε να αποκτήσει τελευταία 20 χρόνια. Απέριψε όμως την πρόσκληση αυτή και μάλιστα είπε ότι δεν εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μολονότι έχει 20 ετή εμπειρία, αυτή περιορίζεται σε συγκεκριμένου τομεί και όχι σε όλου εκείνου τομεί που θα έπρεπε να έχει εμπειρία αν θέλει να εργαστεί ω μηχανικό στη Μάλτα. Επίση, Τα μέτρα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή την επιστολή της 12 η Οκτωβρίου συνάδουν απόλυτα με τις αρμόδιες διατάξεις της οδηγίας. Επίσης, στην επιστολή ο κύριος Μπίλας καλείται να συμμορφωθεί με την σε ρυθμίσεις της Μάλτας που συνάδουν και με την κοινοτική οδηγία. Πρέπει να κάνει περαιτέρω πρακτική άσκηση. Αυτό ζητείται και από την κοινοτική οδηγία και του ζητείται επίσης να περάσει από μία δοκιμασία επάρκειας. Επομένως, τα όσα λέγονται στην επιστολή από τις Μαλτέζικες Αρχές όσον αφορά τα προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχει κανείς για να εξασκεί το επάγγελμα του μηχανικού στη Μάλτα συνάδουν απόλυτα με τις ρυθμίσεις που θέτουμε εμείς στην κοινοτική οδηγία. Επομένως, θεωρούμε ότι η Μάλτα δεν παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Yes, thank you. Uh, I wish to thank the Commission. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολούθησε εκ του στην υπόθεση για να θέσω μια ερώτηση. Ε, σύμφωνα με τι τελευταίε προφορίες που λάβαμε, η Κομισιόν δηλώνει ότι κατά την άποψή οι μαλτεζικέ αρχέ παραβίασαν την οδηγία 2005-36. Θεωρούν ότι εν ώψη των τελευταίων εξελίξεων η Κομισιόν έχει αλλάξει ίσως άποψη περί αυτού. Ναι, η Κομισιόν άλλαξε άποψη διότι εσείς αναφέρεστε στην γραπτή ανακοίνωση που η Κομισιόν υπέβαλε πριν από ένα έτος και πέρυσι υπήρξαν κάποιες εξελίξεις και η σημαντικότερη εξ αυτών ήταν ότι οι μαλτεζικές αρχές αγνόησαν και απέριψαν τα προσόντα λέγοντας στο πρόσωπο ότι δεν μπορείτε να γίνετε δεκτός απλά θα πρέπει να περάσετε κάποια δοκιμασία για την αναγνώριση των προσόντων. Τώρα, η συνεννόηση που υπήρχε ανάμεσα στην Κομισιόν και οκτώ μελών εκπροσώπων της, των μαλτεζικών αρχών επέμειναν ότι έδωσαν την δυνατότητα στον εξεταζόμενο να αποδείξει την επαγγελματική εμπειρία, κάτι το οποίο και συνέβη. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν κατέληξε την 1η Οκτωβρίου ότι τα δικαιώματα του έγιναν σεβαστά, αλλά η απόφαση ήταν πως ο υποψήφιος δεν είχε τα προσόντα που χρειάζονταν Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι ε, συμμορφώθηκε με τον κανονισμό. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ο αναφέρον έπρεπε να έχει την επιλογή ανάμεσα σε μια δοκιμασία επάρκειας, ουσιαστικά μια δοκιμασία που βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και μια ε, περίοδο προσαρμογής, ε, που είναι ουσιαστικά ένα χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί. Αλλά οι συνθήκες που χρησιμοποιούνται τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για αυτή την περίοδο ε, προσαρμογής μοιάζουν πολύ περισσότερο με δοκιμασία επάρκεια τελικά. Δεν είναι τόσο πολύ πραγματική περίοδο προσαρμογής. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω πολύ καλά για ποιο λόγο μία περίοδος προσαρμογής μπορεί να περιέχει στοιχεία τα οποία μοιάζουν περισσότερο με δοκιμασία επάρκεια. Επ' αυτού δεν είμαι ακόμα πεπισμένος με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο αναφέρον είχε την επιλογή και από ό,τι φαίνεται δεν του δόθηκε η επιλογή αυτή από τις αρμόδιες μαλτέζικες αρχές. Θα ήθελα λοιπόν η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανέλθει στο ζήτημα αυτό και να μας πει αν τελικά είναι πλήρως πεπισμένη ότι τα όσα περιγράφονται εδώ πέρα ως περίοδος προσαρμογής είναι πράγματι μία περίοδος προσαρμογής. Ναι, αν έχετε μια διευκρίνηση να κάνετε, σας το λόγο. Ναι. Εγώ δεν μπορώ παρά να επανελάβω αυτά που είπα προηγουμένως. Αυτό βρίσκεται στον ορισμό 3NG για τον ε, περίοδο προσαρμογής. Λέγεται ότι είναι μια περίοδος άσκησης του επαγγέλματος υπό υποπτία και στην επιστολή της 12 Οκτωβρίου λέει ότι ο κύριος ε, Τουλά έχει ένα χρόνο μόνο, θα μπορούσε να έχει κληθεί να κάνει τρία χρόνια, έχει ένα μόνο. Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει ότι ε, ασκείται σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς όπου δεν έχει εκπαιδευτεί και από ό,τι βλέπει πρέπει να κάνει και μια ειδική αξιολόγηση. Αυτό για μας σημαίνει ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την οδηγία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes, well, at this point, Madam Chairman, I... Ναι, πρόεδρε. Θα ήθελα παρακαλώ να παραμείνει ανοιχτό για μία φορά ακόμα μέχρι να έρθω ξανά σε επαφή με τον αναφέροντα και να δω κατά πόσον ικανοποιήθηκε με την απάντηση αυτή. Το θέμα είναι εκδεμές εδώ και πολύ πολύ καιρό. Το να αναβάλουμε άλλη μια φορά δεν είναι τόσο τραγικό. Εάν η κατάσταση πραγματικά είναι ε, ικανοποιητική για τον αναφέροντα όπως είπε η Κομισιόν μπορούμε να το κλείσουμε. Αν συμφωνείτε. Mm, Νομίζω ότι μπορούμε να συμμεριστούμε το έτοιμά σα, διότι έχουν προκύψει κάποιε αμφιβολίε σχετικά με την άποψη που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε αυτή τη φάση της, της πρακτικής άσκησης κλπ φαίνεται πως τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι αυτή η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να ενταχθεί ανάμεσα στις αντισταθμιστικές διαδικασίες που προβλέπουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, ε, όταν δεν υπάρχει αυτοματισμός ε, σε όλη φορά στην αναγνώριση του πτυχίου. Θα πρέπει να παραμείνει λοιπόν ανοιχτό το ζήτημα μετά από ακούσαμε για τον κύριο Μπουζουτήλ θα περιμένουμε περαιτέρω ενημέρωση μετά τι επαφέ που θα έχει. Παραμένει λοιπόν σε κρεμότητα αυτή η αναφορά. Περνάμε στην τελευταία αναφορά της βραδιάς. Αναφορά Μαλτέζου υπηκόου σχετικά με τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2085 από τις αρχές της Μάλτας είναι εκπρόσωπο τη Κομισιόν έχει το λόγο. Ο Κανέλ, ο εκπρόσωπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνοδεύω την κυρία Κανέλ και θα απαντήσω ξενομόλης της Κομισιόν. Να τονίσω πως η οδηγία 2002 85 που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς μετα, ε, μεταφέρθηκε στην ε, Μαλτεζική νομοθεσία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, πρέπει να τονίσουμε. Δεύτερον, ε, θίγεται και το θέμα της ορθής εφαρμογής από πλευράς Μάλτας. Η πρώτη παρατήρηση λοιπόν που θα ήθελα να κάνω είναι πως ε, τα γεγονότα που αναφέρονται αφορούν στο 2007. Τότε η εποχή χρησιμοποιούσε μια διάταξη της οδηγίας που της επέτρεπε να απαλλάξει να απαλλαχθεί από την εφαρμογή της οδηγίας για τα ε, οχήματα στο εθνικό δίκτυο. Από τότε η Κομισιόν δεν έχει λάβει νέα στοιχεία που θα της επιτρέψουν να, ε, να εξετάσει κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή όχι. Πάντως η αναφορά ούτε αυτή περιέχει ικανά στοιχεία για να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αναφέρον και να θεωρήσει πως υπάρχει εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας. Ε, η Κομισιόν εν Ενολίγης δεν έχει στα χέρια της ε, κάποια στοιχεία για να θεωρήσει ότι δεν εφαρμόζεται με τρόπο ορθό η οδηγία. Θα ήθελα λοιπόν ε, περαιτέρω περαιτέρω στοιχεία η Ευρωπαϊκή για να μπορέσει να εξετάσει την διαμαρτυρία αυτή. ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομη. Τι αναφορά δεν αφορά το κατά πόσο έχει μεταφέρει αυτή την οδηγία στο Εθνικό Δίκτυο Μάλτα, αλλά κατά πόσο την εφαρμόζει. Και χαίρομαι που, που η Κομισιόν αναφέρεται στην εφαρμογή της οδηγίας, διότι εδώ στο σημείο που έχουμε η Κομισιόν ε, δείχνει να είναι ικανοποιημένη και με τη μεταφορά της οδηγίας και σταματάει εκεί. Ακούσαμε πως η Κομισιόν έχει προχωρήσει λίγο παραπέρα και εξέτασε την εφαρμογή ακόμα και τώρα, κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι πεπισμένη, ε, για τα όσα μας ανέφερε η Κομισιόν και ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε το, από τον αναφέροντα να μας ενημερώσει αν επισημείνα. να παράσχει περαιτέρω προφορίες για το λόγο τον οποίο αισθάνεται πω η οδηγία δεν εφαρμόζεται επαρκώς. Θεωρώ λοιπόν πως στο σημείο αυτό η αναφορά χρειάζεται να παραμείνει ανοιχτή και ο αναφέρον ε, να του ζητηθεί κατά πόσον κρίνει και για ποιους λόγους ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται. Παναλαμβάνω, δεν πρόκειται για τη μεταφορά της οδηγίας, αλλά για την εφαρμογή της. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις ε, στο έτοιμο του κ. Μπουζουτήλ, θα ζητήσουμε από τον αναφέροντα να μας ενημερώσει περαιτέρω. Ολοκλήρωση της εργασίας μας, εσάβριον.